So, dear colleagues, let's start our meeting with the adoption of the agenda. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίθηκε η μερίσια διάταξη. Έχω μια σειρά ανακοινώσεων. Καταρχήν όσον αφορά ε, μια ενημέρωση για τους ε, τριμερείς διαλόγους. Ο τελευταίος έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου. Εκεί συζητήθηκαν αρκετά θέματα. Ε, η νομισματική προοπτική, το καθεστώς αποκαλύψεων μυστικών, οι κανόνες για τις ε, αρμοδιότητες και επίσης και το γλωσσικό θέμα. Επίσης πρόοδος επιτεύχθηκε για κάποια συγκεκριμένα θέματα. Επίσης η συζήτηση κάλυψε την έγκριση της τεχνικής εργασίας σχετικά με τις ε, προοπτικές, ε, τους παράγονες που πρέπει να αναφέρονται. Αναφέρομαι στην επίσης ανακοίνωση σχετικά με το διαβατήριο και την επόμενη Παρασκευή έχουμε επίσης τριμερή διάλογο στις 7 Νοεμβρίου. Η ανακεφαλαίωση των αποφάσεων των συντονιστών της 24 Νοεμβρίου ε, ο διορισμοί epp διπλή φορολογία, μηχανισμό σε διπλή φορολογία στην Άλντε, ε, η, αξιολόγηση σε θέματα ε, χρεοκοπίας ή το ΕΛΚ, η δυνατότητα ανακεφαλαιοποίησης ε, και αυτό στο ΕΛΚ, η μη ε, απορρόφηση της EBRD και αυτό στο ΕΛΚ, το νέο πακέτο. Εκεί ε, ξακολουθεί και αυτό να είναι κομμάτι του πακέτου, η αναθεώρηση του CRD ε, στην, στους σοσιαλδημοκράτες, cover bond στην ECR, οι καταγγέλλοντες τους πράσινους, η γνωμοδότηση για τη ΣΕΤΑ στο Προεδρείο η γνωμοδότηση για κανόνες ε, περί ε, αφαιρεγγιότητας ε, με αναφορά στον κανόνα 54 στην ΑΛΔΕ. Αυτές είναι οι εκθέσεις που κατακυρώθηκαν. Και για το Brexit μετά από μία σύντομη συζήτηση θα αποφασίστηκε να ακολουθεί και άλλη συζήτηση στις 10 Δεκεμβρίου και κλείθηκε η Γραμματεία να δώσει περισσότερα στοιχεία για θέματα που είναι σημαντικά όπως επίσης και ένα υπόβαθρο για την πολιτική πολιτική ανταγωνισμού. Εξάλλου, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αποφασίστηκε να γίνει άλλη μια συνάντηση στις 4 Δεκεμβρίου. Τα θέματα για την κοινοβουλευτική εβδομάδα ε, του 2017 ε, είναι τα Panama Papers, οι διαρροές τα σταματήματα που μπορούμε να εξάγουμε, Τραπεζική Ένωση, Ένωση Κεφαλαγορών και ε, Νέα Αγορά για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επίσης ε, θα σταλεί μια επιστολή στο, στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Αρχή, θα ζητήσουμε μια ακρόαση και οι συντονιστές ε, συμφώνησαν για το διάλογο να ακολουθήσει αυτός αμέσως ε, μετά το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η οικονομική βοήθεια τεστιά την προσοχή της σε μακροοικονομικά προγράμματα, κυρίως αυτά που αφορούν στην Ελλάδα και όσον αφορά τον έλεγχο των κατεξουσιοδότηση πράξεων, Φεβρουάριος ε, η γραμματεία θα αναζητήσει περισσότερο χρόνο για την οδηγία μύφτη είτε και για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. θα βρείτε και μπορείτε να βρείτε και μια έκθεση με περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν σε αυτή την απόφαση των συντονιστών. Και τέλος, Όσον αφορά στην έκθεση Γκούλα, οι συντονιστές των Πρασίνων ζήτησαν από το ε, Γραμματεία να κάνει μια ανάλυση που να καλύπτει την παράγραφο 19. Οι συντονιστές ε, θα συζητήσουν το επικαιροποιημένο έγγραφο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Είχα πάρα πολλές ανακοινώσεις και τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο σημείο υπαρκών 3 της ημερήσιας διάταξης. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μάρτι Χετεμάκη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής. Είναι ο φορέας εκείνος που όπως γνωρίζετε μπορεί να προσφέρει μια ανεξάρτητη επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος όσον αφορά στον κώδικα ε, ε, διοντολογίας στις ευρωπαϊκές στατιστικές και θέλουμε να συμπεντιμήσουμε το σημαντικό ρόλο που παίζει η έκθεση Σκαπάνο που λάβατε είναι η έκθεση για το στατιστικό αυτοφορέα. Ε, είναι μια έκθεση που έχει σχέση με την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Αυτό είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ. Και θα θυμάστε επίσης ότι είχαμε μία συζήτηση ε, στο πλαίσιο ε, της ομάδας εργασίας με τον κύριο Γεωργίου και με τον κύριο Ράντε Μάκα ναι. και θέλω να υπογραμμίσω ότι το Συμβούλιο αυτό παρακολουθεί εκ του σύναγκες τις συζητήσεις για τον διορισμό του νέου Προέδρου της Eurostat μετά την ε, συνταξιοδότηση του νυν Προέδρου. Αυτά είχα να σας πω ως εισαγωγή και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Χετεμάκη για την ομιλία του. Παρακαλώ, ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την έκθεση του Ευρωπαϊκού Φορέα Στατιστικών Δεδομένων. Η έκθεση αυτή αφορά λοιπόν το ΕΣΚΑΠ, που αποτελείται από έξι μέλη, τον Μάρτιν Κούτσμαν, τελευταίος πρόεδρος της Ισπανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κυρία Κουτσεβονίνη, τέος πρόεδρος της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας και τέος Υπουργό Εργασίας. Πατρίσιο Χάρα, καθηγητής στατιστικών από την Ιρλανδία. Μάριους, Ρουμανία και Κρίτσικοφς που ήταν πρόεδρος της Στατιστικής Υπηρεσίας. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, εξετάζουμε ακόμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα βάσει του κώδικα δοντολογίας, κώδικα πρακτικής. Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε δύο θέματα. Το ένα είναι η πρόκληση εξαιτία των πολλαπλών πηγών πληροφοριών και δεδομένων που χρειάζονται ιδιαίτερη ανάλυση και πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις επίσημες στατιστικές. Ο κώδικας πρακτικής δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως για παράδειγμα το θέμα των πολλαπλών πηγών δεδομένων. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μας έρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές Και τα δεδομένα αυτά φυσικά και πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όμως, πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπου η συγκρισιμότητα είναι κέρια σημασίας. Γι' αυτό το λόγο η ΕΣΚΑΠ προτείνει αξιολόγηση πρώτα των πηγών από όπου μας έρχονται τα δεδομένα και ανάλυση ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά βάσει του κώδικα πρακτικής. Μια δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε έναν επιταχυμένο ρυθμό και να αποφύγουμε να γίνεται κατάχρηση των στατιστικών δεδομένων για πολιτικούς ή άλλους λόγους. Χρειάζονται δεδομένα ποιότητας για να στηρίζουμε και τις πολιτικές αποφάσεις. Τώρα είναι εύκολο online να βρει κανείς ε, πολλά δεδομένα, οπότε είναι εύκολο να καταλήξει σε στατιστικές για να υποστηρίξει κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές δηλώσεις ανεξάρτητα από την ίδια την ποιότητα των δεδομένων. Κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε λαθαμένα μηνύματα ή σε παραπλάνηση. Και το κοινό να αρχίσει έτσι σιγά σιγά να μην έχει εμπιστοσύνη καθόλου στις στατιστικές, ούτε καν τις στατιστικές που προέρχονται από κρατικές αρχές. Συνεπώς πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να έχουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στις ευρωπαϊκές στατιστικές. Συστήνουμε κυρίως οι στατιστικές αρχές να έρχονται σε επαφή πολύ περισσότερο με την κοινωνία των πολιτών για να προωθούν την ε, αξία των επίσημων στατιστικών. Επίσης, οι στατιστικές υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις ε, δημόσιες στατιστικές εφόσον αυτό χρειαστεί. Έρχομαι τώρα στην αξιολόγηση της πρόοδου που έχει επιτευχθεί βάσει του κώδικα πρακτικής. Έχουμε καταλήξει στις διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης. Αναφέρθηκε και ο πρόεδρος λίγο σε αυτά. Οπότε ξέρουμε τώρα πώς θα μπορέσουμε να προσλάβουμε τον νέο διευθυντή της Eurostat και οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περάσουν πια στην νομοθεσία τα κριτήρια επιλογής πρέπει να περιλαμβάνουν την επαγγελματική τους ε, φήμη και την εμπειρία που έχουν στους τομείς που έχουν να κάνουν με την αποστολή του ως επικεφαλής της Eurostat. Η Επίτροπος Τάισεν όλα αυτά τα είπε και τόνισε τον ρόλο της ΕΣΚΑΠ Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τελικά να ακολουθήσει μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής για να ορίσει τον νέο Γενικό Διευθυντή της Eurostat. Αυτή τη χρονιά πάντως υπήρξε καλή πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του κώδικα πρακτικής και τις συστάσεις του peer review. Η συστάση μας είναι η βελτίωση των ε, πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιωθούν και οι ευρωπαϊκές στατιστικές. Θέλω να καταλήξω με το εξή. Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει 16 συστάσεις οι οποίες αναφέρονται στις προκλήσεις πρώτα απ' όλα των πολλαπλών πηγών πληροφοριών, τη σημασία που έχει η εμπιστοσύνη στις στατιστικές και η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του κώδικα πρακτικής ε, στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χετεμέκη, για την παρουσίασή σας. Και έχω πληροφορηθεί ότι με τη διαδικασία επιλογής είσαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με τα θέματα της Eurostat όσον αφορά την επιλογή γενικού διευθυντή. Και όπως επίσης γνωρίζετε, είχαμε εμπλακεί στο πλαίσιο των νέων κανονισμών και σε σχέση και με τον ρόλο του Κοινοβουλίου, σεβόμενη φυσικά την αυτονομή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανεξαρτησία της όσον αφορά εσωτερικά διορισμούς ένα ενδιαφέρον ζήτημα και αυτό. Ερωτώ τους συναδέλφους, υπάρχουν από πλευράς τους ερωτήσεις, παρεμβάσεις, υπερβάνς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στο ζήτημα του ορισμού του διαδόχου, διότι, του πρόεδρου, διότι πρέπει να σταξιδοτηθεί παρόλο που κάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις, κυρίως για ζητήματα που μένα με απασχολούν πολύ, το θέμα της ποιότητας των στατιστικών στον κοινωνικό τομέα, για να έχουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική και την οικονομική πολιτική, αλλά πάση περιπτώσει. Ωραία, τροποποιήθηκε η διαδικασία ορισμού και τα Είπαμε ότι θα συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Καλώς. Εσείς πώς βλέπετε το μέλλον της ε, διεύθυνση και της ανεξαρτησίας της Eurostat, γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται και σε εθνικό επίπεδο. Η Eurostat δεν υπάρχει συνικό τείχος, είναι σύμβουλος της Κομισιόν, έτσι κι αλλιώς η Eurostat. Οπότε συλλέγονται συγκεκριμένα δεδομένα για την κοινωνική πολιτική. Οπότε θέλω να ξέρω ποιος είναι ο ρόλος του δικού σας Συμβουλίου όσον αφορά τη συλλογή και την αναρμόνιση των στατιστικών που παίρνετε από τις χώρες μέλη. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα λοιπόν της ηγεσίας και της ανεξαρτησίας της Eurostat. Ποιες ρήτρες εξασφάλισης έχουμε. Και όταν το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει θα κοιτάξει βέβαια τι θα γίνει με τη διαδοχή του κύριου Ραντρομασέ, του Πρόεδρου, του Διευθυντή, αλλά κατά τη γνώμη σας ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία. Και έρχομαι στη δεύτερη ερώτησή μου που έχει να κάνει με την εξέλιξη του καθεστώτος στατιστικών στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχουμε φτιάξει μια ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα αρρωγής. Είχαμε ανταλλαγέ απόψεων με του υπευθύνου του ελληνικού στατιστικού συστήματος. Είναι ένα ζωτική σημασία στοιχείο για την ε, ανάκαμψη της εμπιστοσύνης. Η Eurostat ε, φυσικά και ενδιαφέρεται όλο ιδιαίτερο. Οπότε εσείς για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Στην επόμενη εσείς ω SGAB Μπορείτε να μας πείτε αυτές τις εξελίξεις πώς τις βλέπετε. Έχετε ένα μήνυμα να μας απευθύνετε για τις εξελίξεις στο ελληνικό στατιστικό σύστημα. Τι πρέπει να γίνει και τι εμείς θα έπρεπε να κάνουμε, θα έπρεπε να εξετάσουμε με κάποιο τρόπο εμείς τα δεδομένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ για αυτές τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις από πλευρά σας. Πρώτον, όσον αφορά την ανεξαρτησία της Eurostat. Συζητήθηκε αυτό διαμακρών όταν είχαμε την πρώτη ελληνική στατιστική κρίση και υπήρχαν και διαφορετικές προτάσεις για την αλλαγή του καθεστώτος της Eurostat. Και τέλος, η τελική λύση ήταν ότι θα υπήρχαν περισσότεροι έλεγχοι για την ε, ισορροπία και αποτελεσματικότητα της Eurostat και πολύ σημαντικός ήταν ο τροποποιημένος κανονισμός ε, 2-3, όπου το Κοινοβούλιο είχε ένα σημαντικό ρολό να διαδραματίσει σε αυτό το πλαίσιο. Παρότι οι διαδικασίες επιλογής δεν είχαν κατοχυρωθεί νομικά, η ιδέα επιλογής του Γενικού Διευθυντή της Eurostat με βάση αντικειμενικά κριτήρια και ικανότητες και δεξιότητες ε, ειδικά σε σχέση με τη Eurostat ε, ήταν δεδομένα ως στοιχεία και αυτό έδωσε και σε μένα την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ήταν ο στόχος του νέου αυτού κανονισμού να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί και δίνει συνέχεια σε αυτή τη διεργασία, σε αυτές τις διεργασίες σε αυτή τη διαδικασία που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον νέο κανονισμό και διέπεται από αυτόν σε σχέση και με ένα νομικό πλαίσιο. Δεύτερον, τότε υπήρχε και μία πρόταση ως λύση να δημιουργηθεί η ΕΣΚΑΠ και η ΕΣΚΑΠ δηλαδή ακριβώς ο Ευρωπαϊκός Συμβουλευτικός Φορέας για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής όσον αφορά την εποπτεία και των εθνικών ε, ε, στατιστικών υπηρεσιών και της Eurostat επικουρικά ιδιαίτερα. Και τώρα θα έλεγα ότι έχουμε ένα αρκετά καλά ισορροπο, ισορροπημένο σύστημα με ελέγχους ε, και ισορροπίες για το πώς δηλαδή συνολικά λειτουργεί και διαδραματίζει το ρόλο της ε, ε, η ΕΣΓΑΠ ως ε, στατιστικός φορέας, στατιστικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη πλευρά επίσης πρέπει να το πω αυτό ότι όταν συζητήθηκε η αναθεώρηση, η μεταρρύθμιση, ήταν σαφές ότι οι στατιστικές υπηρεσίες ούτε στα κράτη-μέλη, αλλά ούτε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να είναι απόλυτα ανεξάρτητες αυτές οι υπηρεσίες όπως είναι ανεξάρτητες οι κεντρικές τράπεζες. Πάντα αποτελούν μέρος και τμήμα της κρατικής διοίκησης, της κρατικής δομής διοίκησης. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει κανείς είναι να δημιουργηθούν όροι και προϋποθέσεις ώστε με αυτά τα προαπαιτούμενα να διασφαλίζεται η επαγγελματική επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Ιδρύματος σε περίπτωση ε, της Eurostat για παράδειγμα. Έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα για την Ελλάδα. Ποια είναι η άποψη της ΕΣΓΑΠ. Τώρα φυσικά εκδώσαμε αρκετές γνωμοδοτήσεις όσον αφορά τα θέματα ελληνικής στατιστικής, Greek statistics, και υπήρξαν και θετικές εξελίξεις από την άλλη πλευρά όμως είχαμε μετά και την επανεμφάνιση νομικών διαδικασιών κατά του πρώην Προέδρου και ε, συναδέλφων του. Και φυσικά όλα αυτά, αυτές οι προσφυγές και διαδικασίες οι νομικές βασίστηκαν σε εικαζόμενη, εσφαλμένη διαβίβαση στοιχείων που συνεπαγόταν ε, και το επίπεδο της Eurostat και τις ε, επίσημες απαιτήσει για αυτά. Και με ιδιαίτερη ανησυχία είδαμε την επανεμφάνιση αυτών των νομικών διαδικασιών και προσφυγών εις βάρος του πρώην Προέδρου της ε, ελληνικής ε, εθνικής στατιστικής υπηρεσίας και κατά δύο συναδέλφων του επίσης. Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να πράξει η δική σας κοινοβουλευτική επιτροπή και τι μπορούμε να πράξουμε εμείς. Θα έλεγα αυτό το οποίο πράξατε ήδη μέχρι τούδε είναι πολύ σημαντικό. Είχατε τις ακροάσεις και τη συζήτηση, τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν με τον πρώην πρόεδρο της ε, Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και με τον κύριο Ράδερμαχερ επίσης. Και δόθηκε δημοσιότητα σε αυτό το ζήτημα και από πλευρά σας. Είναι η ήπια δύναμη και η, το δυναμικό αυτής της ήπιας εξουσίας που έχουν τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα στη διάθεσή τους να παρεμβαίνουν με τέτοιο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενημερώνονται όλοι για το ποιο ήταν το σκηνικό και το τοπίο και η προϊστορία όσον αφορά αυτή την υπόθεση και ποια είναι τα αντικειμενικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων αυτή μαζί σας και είναι και στο διαδίκτυο μεταδίδεται επίσης. Και, έχουμε και υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις από πλευράς μου. Πρώτον, αναφερθήκατε σε έναν αριθμό σημαντικών νομοθετικών βελτιώσεων όσον αφορά το ευρωπαϊκό στατιστικό πλαίσιο και τον δεοντολογικό κώδικα και τον κανονισμό 223. Θα λέγατε, πιστεύετε ότι βρισκόμαστε τώρα στην φάση της υλοποίησης και εφαρμογής ή θεωρείτε ότι και κάτι άλλο θα έπρεπε να προσθεθεί ως βελτίωση, αλλαγή πλαισίου αυτού του πλαισίου ή του δεοντολογικού κώδικα ή του προϋπολογισμού ή κάποιων πρόσθετων στοιχείων όσον αφορά αυτό το καθεστώς. Δεύτερη ερώτηση αφορά, γιατί κάνατε εσείς αυτή την αναφορά σε, στην παρέμβασή σας για την, το πλαίσιο, το κλίμα μετά τις πολιτικές παρεμβάσεις όσον αφορά τη στατιστική και για την ε, από πολιτικής πολλάκης κατάχρηση ίσως αυτών ε, των στοιχείων. Πώς βλέπετε εσείς ότι θα έπρεπε να διαμορφωθεί αυτός ο ρόλος, πώς θα μπορούσε να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί μέσα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ισορροπία ακριβώς σε σχέση με αυτά τα στοιχεία ώστε να αποφεύγονται καταχρήσεις. Και τέλος φυσικά είσαστε ελεύθερος να σχολιάσετε ή να μην σχολιάσετε τη συγκεκριμένη ερώτηση για κάποιους από τους δείκτες που βρίσκονται υπό συζήτηση και εξέταση και μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο όσον αφορά την στατιστική παράμετρο φυσικά εδώ για τα οικονομικά γίνεται μια συζήτηση για την απλούστευση όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες και κανονισμούς και υπάρχουν ευρύτερες συζητήσεις στο Συμβούλιο που αφορούν το πώς κάποιοι από τους δείκτες αυτούς μπορούν να καθοριστούν ιδιαίτερα σε σχέση με μια δομή, πώς όλα αυτά διαμορφώνονται διάβασα ενδιαφέροντα σχόλια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναφέρθηκε ότι δεν χρησιμοποιείται αυτός, δεν χρησιμοποιούνται τέτοιοι δείκτες διότι μπορούν να τύχουν πολλών ε, ερμηνεών. Από την άλλη πλευρά όμως είναι ένας από τους πυλώνες ε, το καθεστώς αυτών των δικτών ε, για τα στατιστικά. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το αξιολογείτε. Σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θίγεται. Πρώτο ζήτημα, αν το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν επαρκεί ή όχι. Ναι, θα έλεγα επαρκεί, είναι επαρκές. Υπάρχει μια καλή ισορροπία πραγμάτων όσον αφορά τις νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσει. Από την άλλη πλευρά όμως όσον αφορά τον δεοντολογικό κώδικα, τον κώδικα πρακτικής, το Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΓΑ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να επικαιροποιείται αυτός ο κώδικας πρακτικής, διότι οι νέες προκλήσεις που προέρχονται από τις πολλαπλές πηγές ε, στοιχείων και των big data μεγάλων δεδομένων μεγάλων διαστάσεων δεδομένων και το πώς χρησιμοποιούνται αυτά ή μπορούν να χρησιμοποιούνται ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα για να είναι αξιόπιστα αυτά τα στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη. Να είναι μετρήσιμα και συγκρίσιμα. Είναι πρόκληση για όλες τις στατιστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να έχουμε να επιτύχουμε κάποια συμφωνία, πώς θα χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία. Διότι πάρα πολλές από τις πολιτικές μας εξαρτώνται από τη συγκρισιμότητα αυτών των στοιχείων. Δεύτερα, δεύτερον, ερωτήσατε στην παρέμβασή σας για την μετά την πολιτική παρέμβαση περίοδο ή φάση και τι θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με αυτό το θέμα. Φυσικά οι υπεύθυνοι για τα, τη, στα, τη στατιστική ως προς αυτό το θέμα πρέπει να θεωρήσουμε ότι εμπλέκονται ένα παράδειγμα να αναφέρω στην αναθεώρηση των στοιχείων για το ΑΕΠ από πλευράς Ιρλανδίας νωρίτερα εφέτος, η αύξηση του ΑΕΠ της Ιρλανδίας για το 2015 αναθεωρήθηκε στο 26,3%. Και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό, αυτή η επικαιροποίηση, αναθεώρηση. Είναι σαφές ότι και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο εθνικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερα στοιχεία νωρίτερα που να δικαιολογούν και να επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους ή κατέστη αναγκαίο να γίνει αυτό. Και μετά, έπειτα, αν μόνο αυτά τα γεγονότα, τα στοιχεία αναφέρονται χωρίς κάποια επεξήγηση, τότε ίσως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το ότι δεν δείχνουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στα επίσημα στατιστικά στοιχεία πολυπολίτες Και ίσως εδώ μπορεί να υπάρχει και κάποια ουσία που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση. Οι δημοσιογράφοι για παράδειγμα επιθυμούν και χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για τέτοιου είδους ε, στατιστικά δεδομένα. Και πρέπει να δούμε για το πώς γίνεται αυτή η επιλογή στοιχείων και η ε, διήλυση στοιχείων θα πρέπει να μπορεί να διευρύνει κανείς την κατανόηση των στατιστικών αυτών στοιχείων και δεδομένων και να μπορεί να κατανοήσει το ότι υπάρχει ανάγκη να θεωρούν αξιόπιστα τα στατιστικά αυτά στοιχεία οι πολίτες. Και δυστυχώς η εμπιστοσύνη αυτή όσον αφορά αυτή την αξιοπιστία από πράγμα πολιτών δεν βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα ήταν ευκταίο και επιθυμητό και αυτό αποβαίνει εις βάρος των ευρωπαϊκών πολιτικών διότι πάρα πολλές από τις πολιτικές μας βασίζουν ακριβώς σε στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία σας ερώτηση. Κάνατε μία ερώτηση για τους δείκτες στην παρέμβασή σας και όσον αφορά και την, το θέμα του ε, ελίμα και αν επιτρέπετε να σχολιάσω παρότι αυτό δεν βρίσκεται στην άμεση εντολή της ΕΣΚΑΠ ως ε, ε, αρμοδιότητα υπάρχει μια σαφής λογική των πραγμάτων όταν χρησιμοποιεί κανείς τέτοιου είδους συντελεστές και δείκτες ε, για τα ελλείμματα, διαφορετικά ελλείμματα. Και πρέπει να αντιμετωπίζετε επίσης να λαμβάνετε υπόψη και η κυκλική εξέλιξη πραγμάτων στα δημοσιονομικά μιας χώρας. Και γι' αυτό είναι πολύ θετική η ε, θα έλεγα ε, τεκμηρίωση στην χρήση των διαρθρωτικών ελλημάτων στις δράσεις μας. Οι κανόνες φυσικά βασίζονται πολλαπλά στις ε, συστάσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαθροτικών ελλημάτων. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο καθιστά επιτακτική την ανάγκη χρήσης αυτών των δικτών και στοιχείων για την μέτρηση αυτής της κατάστασης. Το γεγονό ότι είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς κάτι δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόσχημα εδώ η δικαιολογία για να ακολουθούνται αρνητικές, μη θετικές, κακές πολιτικές. Και αν δει κανεί τι ελλείψεις που υπάρχουν πολλές φορές, τότε θα πρέπει να βελτιώνονται τα πράγματα και όχι να δικαιολογούνται τα κακοσκήμενα και να προσπαθούμε να υπερβούμε αυτές τις ε, ελλείψεις ε, και ανεπάρκειες. Εξάλλου υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι που ακολουθούνται παγκόσμια όσον αφορά την μέτρηση των θωτικών ελλημάτων. Για παράδειγμα, όσον αφορά το CBO, Congressional Budget Office, ε, στις ΗΠΑ, έχω μια δεδομένη ε, προτίμηση σε σχέση με τις μεθόδους που ακολουθούμε και χρησιμοποιούμε από πλευράς Ευρώπης. Αυτό που θα ήθελα να πω όμω είναι, είναι ότι υπάρχει ε, μια δυνατότητα μεθοδολογικού μείγματος policy mix στο mix κατά τη μέτρηση αυτών των πραγμάτων που θα μπορούσε να ήταν θετικό για το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστούμε και εμείς. Αν δεν υπάρχει ε, κάποια άλλη ερώτηση, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για την πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία που μας προσφέρατε και ήρθατε εδώ και θα παραμείνουμε σε στενή επαφή και σε διάλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.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 Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο υπερθμών 4 της ημερήσιας διάταξης ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017. Ο συγητής είναι ο κύριος Χοκμάκ, ε, ο οποίος έχει καταθέσει το σχέδιο της έκθεσής του. Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συζητήσεις ε, που είχαμε μέχρι τώρα σχετικά με την ε, ετήσια ανάπτυξη, επισκόψη της ετήσια ανάπτυξης. Ε, αυτό το έγγραφο της Κομισιόν και το δικό μου το έγγραφο είναι πραγματικά πολύ σημαντικά γιατί αυτά καθορίζουν τα πλαίσια για τις συζητήσεις αλλά και για τις ε, πολιτικές δράσεις. Επίσης και καθορίζουν και για το πλαίσιο για το πώς πρόκειται να προσανατολιστεί η Κομισιόν εφαρμόζοντας τις ε, πολιτικές και τους κανόνες. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ανάπτυξη ανακάμπτουμε με αργό ρυθμό, αλλά ανακάμπτουμε. Και επίσης όλα αυτά κατέστησαν δυνατά από μια πάρα πολύ δαπανηρή νομισματική πολιτική, η οποία όμως δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είναι μια νομισματική πολιτική η οποία όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΚΤ, ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί στο δίνεκες γιατί ε, περικλεί σε τελική ανάλυση και ε, νομισματικούς και χρηματοψητικούς κινδύνους. Άρα δηλαδή η ανάπτυξη είναι εύθραυστη. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούν να καθιστούν την ανάπτυξη βιώσιμη, μακροπρόθεσμα, αλλά και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και επ' αυτού νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας. Μέχρι εκεί συμφωνούμε όλοι. Και κατόπιν περνάμε στη συζήτηση σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε πιο ευέλικτη στάση. Και νομίζω αυτό θα είναι το επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων. Αλλά επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω το εξή. Σε περιόδους ανασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην υπονομεύουμε τις ε, προϋποθέσεις για τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυτή η σταθερότητα συμβαδίζει με το σύμφωνο σταθερότητας γιατί αν υπάρχει ανασφάλεια σχετικά με το σύμφωνο αυτό τότε δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομία και θέλω να υπογραμμίσω κύριε Πρόεδρε ότι δεν θέλουμε κι άλλες ανασφάλειες στην ευρωπαϊκή οικονομία ρίχνοντας ε, μια ματιά τριγύρω είναι καθίσατε σαφές ε, ότι το σύμφωνο ε, σταθερότητας ε, ενισχύει την οικονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι αν αμφισβητήσουμε το σύμφωνο σταθερότητας με την νομοθεσία που έχουμε υφίσταται κίνδυνος να υπονομεύσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη σταθερότητα από τις επενδύσεις. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα στο πρόσφατο παρελθόν και θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν ε, ότι τα ελλείμματα δεν ε, είναι ένα ψημά για την ανάπτυξη των αντίον δημιουργούν μεγαλύτερα ελλείμματα, μεγαλύτερα βάρη και μεγαλύτερες ανασφάλειες. Αν υπήρχε μία λύση ε, για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, δηλαδή να ε, θερμαίνεται, να αναθερμαίνεται η οικονομία με ελλείμματα, τότε θα τα αφήναμε να αυξάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Εκείνο που είναι σίγουρο ότι στις ευρωπαϊκές οικονομίες δεν μας λείπουν τα ελλείμματα. Αυτό όμως που διαπιστώσαμε είναι ότι τα ελλείμματα προκαλούν μεγαλύτερα βάρη, μεγαλύτερο ε, κόστος ε, των τόκων, λιγότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και ε, ε, οδηγούν σε μακροπρόθεσμη έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Όσο πιο πολύ ακολουθούμε αυτό το δρόμο, τόσο περισσότερο υπονομεύουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ανοίξουμε μια ματιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και έχουν εξηγιάνει τα δημόσια οικονομικά τους, έχουν ε, δει να προκύπτουν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία να ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο. Αν δεν το κάνουμε θα αντιμετωπίσουμε όλο και μεγαλύτερα προβλήματα. Γνωρίζω μερικοί συνάδελφοι λένε ότι με ελλείμματα μπορούμε να σταματήσουμε τη λιτότητα. Το αντίθετο ισχύει κύριε Πρόεδρε. Σε χώρες όπου τα ελλείμματα διωγγώνται συνεχώς, στο τέλος επιβάλλεται δρακόντια λιτότητα. Όμως στα κράτη-μέλη όπου έχει υπάρξει ε, δημοσιονομική εξυγίανση και έχει δημιουργηθεί και μια σταθερή πλατφόρμα για επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα. Εμείς λοιπόν η δική μας ευθύνη είναι να επιδιώκουμε την ανάπτυξη γιατί αλλιώς ε, η λιτότητα θα είναι το συνεπακόλουθο των όλο μεγαλύτερων ελλημάτων. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Από νομική ε, σκοπιά υπάρχουν οι κανόνες και είναι καθήκον της Επιτροπής να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Δεν είναι δουλειά της Επιτροπής να αλλάζει τους κανόνες που έχουμε, αλλά η δουλειά της Κομισιόν είναι να εφαρμόζει τους κανόνες. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νομική ένωση Πιστεύω λοιπόν ότι ε, πρέπει να μπούμε σε μία συζήτηση για πιο ε, ποιοτικά δημοσιονομικά. Κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τόσοι πολλοί θεωρούν ότι οι σημαντικότερες ε, δαπάνες θα πρέπει να είναι περισσότερο ή κάτω από το 3%. Εγώ πιστεύω ότι οι σημαντικότερες δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στο 100% των εσόδων των κρατών μελών. Και όταν αλλάζουν τα πράγματα δεν μπορεί να ισχύει το μείον τρία. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί οι εγγραφές των προπολογισμών γίνονται αντίστροφα. Δηλαδή οι πιο σημαντικές δαπάνες είναι τελικά το επιχείρημα για να αυξηθούν τα ελλείμματα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία και να δείξουμε υπευθυνότητα όχι μόνο για να σεβόμαστε τους κανόνες αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις και εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι για μένα και για τη δική μου την πολιτική ομάδα είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν θα λειτουργήσει ως θεματοφύλακας των συνθήκων και της κείμενης νομοθεσίας. Προσβλέπω λοιπόν στις συζητήσεις με τους και ηγητές προφανώς πρέπει να συζητήσουμε. Ε, για να το πω έτσι, το λιγότερο μπορώ να πω είναι, είναι, σαφές ότι μας χωρίζουν πράγματα εδώ, στο Κοινοβούλιο, αλλά οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας επί της οποίας έχουμε αποφασίσει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδες εισηγητές. Πρώτον, από τους σοσιαλιστές, Πέτρο Σίλβα Περίγρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή για τα σχόλιά του. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα συνεργαστούμε προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Παρόλο που συμφωνώ ότι μας μένει πολλή δουλειά ακόμα, αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και σε συμβιβασμούς. Γι' αυτό, γιατί όπως είπε και ο συγκεκριτής, έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά αυτά τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Πάντως πιστεύω ότι είναι εφικτό. Έγινε και στο παρελθόν, οπότε δεν μπορώ παρά να ελπίσω ότι θα συνεργαστούμε καλά για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν όσον αφορά την κατάσταση. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε για το ότι υπάρχει ανάκαμψη, η οποία όμως είναι εύθραυστη, και ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα αποκλήσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, όλος ιδιαίτερος. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Ωραία, έχουμε κάνει εκθέσεις και κατά το παρελθόν, έχουμε ζητήσει επενδύσεις για την ανάκαμψη, σύγκληση. Οι τίτλοι είναι πάντα ξεκάθαροι. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπατε κι εσείς, δεν μας λέει ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να συμπληρωθεί από άλλες πολιτικές, δημοσιονομικές, φορολογικές, διαρθρωτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μας λέει κάτι παραπάνω. Τώρα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα τα εργαλεία, νομισματικά, δημοσιονομικά, φορολογικά κτλ. πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τώρα υπογραμμίζονται οι άλλες πολιτικές, εκτός από την νομισματική δηλαδή, για να διασφαλίσουμε την οικονομική ανάκαμψη. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα λέει ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες δημοσιονομικές πολιτικές. Αυτό είναι κάπως καινούριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εδώ το συζητάμε εδώ και καιρό. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει ε, περισσότερο να συμμετέχει η δημοσιονομική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα. Η πρόταση λοιπόν τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παίρνει τη μορφή μιας συγκεκριμένης πρότασης. Positive Fiscal Stance το λέει. Δηλαδή θετική δημοσιονομική πολιτική για το 0,5% του ΕΠ. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πρόταση και είναι μια πολιτική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το πρώτο που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι Ποια είναι η πολιτική απάντηση που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την πρόταση. Βλέπω ότι εσείς προτείνετε να πούμε σημειώνουμε την πρόταση. Εντάξει, λαμβάνουμε γνώση. Ωραία, εγώ θα ήθελα κάτι κάπως πιο θετικό για αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα που έχουμε, αν θέλουμε επενδύσεις. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, τότε βεβαίως και πρέπει να έχουμε μια περισσότερο θετική συνεισφορά στη δημοσιονομική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας ζητάει να παρετηθούμε από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν είναι εδώ πέρα από την πράγμα διαλέξουμε ύφεση ανάπτυξη. Όχι βέβαια. γνωρίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα για τα δημόσια οικονομικά με επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη. Η λιτότητα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μερικές φορές αντί για αποτελέσματα. Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο είναι να συζητήσει την πρόταση αυτή. Να την δει, να μην την αγνοήσει, να την εξετάσει και να τοποθετηθεί πολιτικά επ' αυτής. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι βεβαίως και καταλαβαίνω όλη τη συζήτηση που γίνεται για την αξιοπιστία των κανόνων. Αλλά εγώ δεν βλέπω γιατί πρέπει να κάνουμε μια στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία για το υπερβολικό έλλειμμα. Αυτή είναι μια συζήτηση που παραπέμπει στο όσο έχουμε συζητήσει για την Ισπανία και την Πορτογαλία πρόσφατα. αποφασίσαμε και καλά κάναμε να μην επιβληθούν κυρώσει στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Συνεπώς, αυτά πιστεύει η ομάδα μου και θέλω να προσθέσω και δύο ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι χρειάζονται επενδύσεις. Και σίγουρα το γνωρίζετε κι εσείς αυτό ο συζητητής. Όμως η μνήμα στις επενδύσεις εδώ συνδέεται και με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τις Επενδύσεις της Κομισιόν. Και σίγουρα θα θέλει να το παρατείνει η Κομισιόν και πρέπει να υπάρξει σαφής τοποθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού. Και τέλος, τα κοινωνικά προβλήματα και σύγκληση. Εδώ νομίζω ότι το μήνυμά μας επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για την ανάκαμψη. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αποκλίσεις που σκοτώνουν τις προσπάθειές μας. Κατόπιν τούτων, επαναλαμβάνω ότι πιστεύω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό προσβλέπω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Για την ίσια, Ρόμπερτ Ζήλε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με ευχαριστίες σε σχέση με τον εισηγητή και για την αρχική παρέμβαση του Γκούναρ Χεκμάσκ. Και φυσικά δεν είναι οι ίδιες οι απόψεις ε, ευρύτερα στο σώμα. Η ανάλυση σωστά ταυτοποιεί τα περισσότερα προβλήματα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υψηλό ποσοστό μη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και η μεγάλη ανάγκη των μεταρρυθμίσεων σε κάποια κράτη-μέλη που δημιουργούν γενικά ένα πολιτικό κλίμα που υφίσταται γύρω από αυτό το πρόβλημα. Επίσης για τους κινδύνους όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν τα θεσμικά όργανα ε, και να συμμορφώνονται με κανόνες ε, και όχι τόσο να δημιουργούν διαρκώς κανόνες. Υφίστανται μη ισορροπές σχέσεις ε, και το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι το ζήτημα των πλεονασμάτων έναντι των ελλημάτων. Ενώ διαρκώς πολλοί Μελετητές και επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι είναι ένας από τους κύριους συντελεστές όσον αφορά τη μη ισορροπή κατάσταση στην ε, Ευρωζώνη. Θα πρέπει να σημειωθεί και όπως σωστά αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες χώρες με υψηλά ελλείμματα έχουν επιτύχει κάποιες προόδους όμως σε πολλές άλλες ε, ε, περιπτώσεις και σε ανεπτυγμένες χώρες όπως στη Γερμανία συνεχίζει να αυξάνεται και είναι θετικό το να καλύπτεται από την έκθεση αυτή η πτυχή πριν από κάποια χρόνια σε σχέση με τους Υπουργούς Οικονομικών, σε σχέση με την σύγκριση και την ε, σύγκριση όσον αφορά και ε, τα ποδοσφαιρικά, ακόμα και όταν υπάρχουν καλές ε, επιδόσεις, βλέπει κανείς ότι πολλές φορές ε, οι ε, φύλαθλοι όταν δεν έχουν ενδιαφέρον και μπορεί να ε, κριθεί το αποτέλεσμα εκ των προτέρων δημιουργούνται προβλήματα για το άθλημα και σε σχέση με τις μη ισόρροπες σχέσεις οικονομικά πρέπει να αντιμετωπιστούν διότι δημιουργείται πρόβλημα διαφορετικά και θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, ξεπεράσουμε το προεμένος Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει το σωστό είδος επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αν υπάρχουν προγράμματα επενδύσεων ε, σχετικά και με την πρικοδότηση αυτών των σχεδίων δεν μπορούμε να έχουμε σοβαρά αποτελέσματα σε σχέση με τις ε, επενδύσεις ε, κινδύνου που προσπαθεί κανείς να προσελκύσει σε μια χώρα έναντι του τι συμβαίνει από πλευράς ε, κρατικών αρχών. Αν χρησιμοποιούμε ως δημόσιο μέσο αυτά τα προγράμματα και ταμεία, αυτά τα σχέδια και ταμεία θα πρέπει να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεβασμό για μια πιο ισόρροπη, ελελογισμένη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Για την Άντε Βιετνίκ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Βιερίνκ. Θέλω να ευχαριστήσω για το σχέδιο έκθεσης στον εισηγητή. Με ικανοποιεί το ότι ο εισηγητής το περιεχόμενο αυτό το ε, κρατά σε ένα ε, πλαίσιο το οποίο ε, σε σχέση με την ετήσια ανάπτυξη ακολουθεί την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη στρατηγική του τριγώνου επενδύσεων όσον αφορά μια υπεύθυνη δράση. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία που έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για μας. Η σπουδαιότητα στις επενδύσεις στη γνώση, στην έρευνα, ανάπτυξη, στις επιστήμες που θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα για τη δημιουργή θέσης απασχόλησης. Έχουμε μια ευκαιρία να γίνει αυτό το, κύριο, ε, το πιο δυνατό μας χαρτί όταν ανταγωνιζόμαστε άλλες χώρες. Αυτό απαιτεί λοιπόν να γίνουν επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και από τους ε, ιδιώτες επενδυτές. Είναι σημαντική αυτή η πρόσβαση ιδιαίτερα για επιχειρήσεις ε, που ακολουθούν μια πολιτική έκθεση σε κινδύνους. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην προσπελασιμότητα στις επενδύσεις. Πολλές φορές ε, οι αγορές δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Πρέπει να πετύχουμε μια πιο ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία της Κεφαλαιακής Ένωσης. Ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ε, πανευρωπαϊκά σχέδια και μέτρα μέσω των επενδύσεων. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να απελευθερωθούν επενδύσεις όπου χρειάζονται περισσότερο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει να ε, επενδύσει σε διασυνοριακές επενδύσεις, στην καινοτομία, στην γνώση, στα ψηφιακά. Και στις, ε, θεωρούμε ε, ότι εδώ υπάρχουν ελλείψεις και πρέπει να καλυφθούν. Το ΕΦΣΥ θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνο ένα θέμα του πώς μπορούμε να την αυξήσουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα, είναι επίσης ζήτημα του πώς μπορούμε να επιτύχουμε τον θεμητό ανταγωνισμό. Το dumping είναι εκείνο το οποίο ζημιώνει και την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την, τον αθέμητο ανταγωνισμό ταυτόχρονα ενώ προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας γιατί διαφορετικά προσπαθεί κανείς να εκαθαρίσει μια κατάσταση ενώ διαρκώς δημιουργούνται προβλήματα. Ο εισηγητής έχει κάνει μια σειρά σημαντικών προτάσεων. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ως θεματοφύλακας των συνθήκων χωρίς αυτήν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα απολέσει την αξιοπιστία του. Ο εισηγητής σωστά αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προσέχουν και την ποιότητα των προϋπολογισμών τους και πραγματικά αυτό έχει επιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά και ευφιέστερα στην κατάρτιση και χρήση των προϋπολογισμών τους πρέπει να μπορούν από την κατανάλωση να δημιουργούνται πόροι, να μετατίθενται από την κατανάλωση στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης. Τώρα για τα το φορολογικό και για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών. Πρέπει να αξιολογηθούν πολύ προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητής σωστά τονίζουν τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αφορμή τις δημογραφικές αλλαγές. Θα έχουμε όλο και έναν πιο υπερήλικα πληθυσμό που θα πρέπει να φροντίζουμε. Οι άνθρωποι θα ζουν περισσότερο θα πρέπει λοιπόν εδώ αυτά τα πλήγματα, τα δημογραφικά εντός εισαγωγικών να αντιμετωπιστούν όσον αφορά τις συντάξεις για παράδειγμα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές ευθύνες ε, για τις, τις συντάξεις και την ε, σύνδεση και την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους. Έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιος είναι ο πραγματικός χώρος που μπορούμε να καλύψουμε στην Ευρώπη με τις δράσεις μας. Υποστηρίζουμε γενικά λοιπόν την, το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή με κάποιες προσθήκες και τροπολογίες. Ευχαριστώ. Μιγγέλ Βιέγας από την ΚΟΕ τώρα, παρακαλώ. Mm. Καλό σας απόγευμα. Σημειώνω ότι αυτό το οποίο αναφέρθηκε και με την ε, ανησυχία ότι έχουμε εδώ ταυτολογίες όσον αφορά κάποιες αλήθειες για το ότι δηλαδή τα ελλείμματα δημιουργούν και ζήτημα στην υπερχρέωση. Αυτό είναι εκ του περισσού. Όμως ε, το κυριότερο θέμα, ε, μια και κανείς δεν θέλει να δημιουργούν ελλείμματα χάρη ελλειμμάτων το θέμα το οποίο τίθεται είναι σε μια κρίση, κρίση οικονομική, πρέπει ή όχι οι κυβερνήσεις ε, να δημιουργούν κάποια ελλείμματα ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποια κίνητρα για την ε, ανάπτυξη και να μπορέσει η οικονομία να ανακάμψει. Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. Κανένας δεν θέλει να υπάρχουν ε, ελλείμματα ως ελλείμματα. Όσον αφορά την αξιοπιστία τώρα, εγώ συμφωνώ με αυτή την ιδέα του ότι δηλαδή πρέπει πραγματικά να είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερης εμβέλειας σήμερα. Η κρίση αξιοπιστίας όσον αφορά και το ευρώ και όλου του οικοδομήματος με κανονισμούς, οδηγίες κτλ δεν απορρέει από μεμονωμένη στάση κάποιας χώρας, αλλά από την ίδια την πραγματικότητα της ε, εφαρμογής των κανόνων και κανονισμών από ευθύς εξ αρχής από την δημιουργία του ευρώ. Και ευθύ εξ αρχή από την δημιουργία του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη με του ε, κανόνε και κανονισμού που εφαρμόζονται σε κάποιε χώρες αλλά όχι σε κάποιε άλλε. Με την κατάργηση αυτή τη συμφωνία το 2004 από τη Γερμανία και Γαλλία με μια λιτότητα αντιπαραγωγική που δεν καταλαβαίνουν και δεν δέχονται οι πολίτες. Δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι αναγκαίο εξ ονόματος της διάσωσης ενός οικονομικού συστήματος να δημιουργηθούν προγράμματα περικοπών και λιτότητας που δεν επιλύουν τα προβλήματα. Και για αυτούς τους λόγους αυτό είναι στην ουσία το ζήτημα λοιπόν. Και έχουμε ένα παράδοξο εδώ, έτσι δεν είναι. Με άλλα λόγια, η πορτογαλική κατάσταση θα έπρεπε να αξίζει κάποιον αναστοχασμό που είναι καρπός ε, δυνάμεων που απέρευσαν από τις εκλογές του Οκτωβρίου πέρυσι και ουσιαστικά κυρώνονται μέτρα στο σύνολό τους που επιβλήθηκαν από την Τρόικα. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται σε σχέση με τις συμβάσεις. Ε, τις ώρες απασχόλησης, ε, για την ε, ε, αύξηση των εσόδων, την ελάφρυνση φόρων και επιβαρύνσεων και την σπάυση προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης και παρόλους τους κινδύνους και απειλές που υπάρχουν και παρότι υπάρχουν διαρκείς πιέσεις που ασκούνται και σύμφωνα με τις οποίες θα καταβυθιζόταν και θα καταστρεφόταν η Πορτογαλία, όχι μόνο δεν καταβυθίστηκε και δεν καταστράφηκε, αλλά συνεχίζεται η οικονομική της ανάπτυξη. Ο, και η ίδια όσον αφορά την δημοσιονομική κατάσταση δείχνει μια βελτίωση όσον αφορά το έλλειμμα και όλα αυτά θα έπρεπε να αξίζουν από πλευράς μας έναν αναστοχασμό, ένα προβληματισμό σε σχέση με τα θέσφατα αυτού του δόγματος για την ε, λιτότητα. Διότι αυτά τα οποία συζητούμε εμείς ε, έγκυνται σε μια ερμηνεία φονταμενταλιστική των κανόνων και κανονισμών της επιτακτικής λέει ανάγκης ε, για μια πολιτική λιτότητας αγνοώντας την ουσία αυτό που είναι οι συνέπειες και τα ίδια τα αποτελέσματα της εφαρμογής των κανόνων ε, του ευρώ που στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών των χωρών δεν έγιναν ποτέ κατανοητοί αυτοί οι κανόνες και συνεχίζουν να ακολουθούν τα ίδια, τους, τις ίδιες πολιτικές με το ίδιο πληκτρολόγιο σε σχέση με την λέει ανάκαμψη των επενδύσεων. Και στην Πορτογαλία βρισκόμαστε ενώπιον μιας πτώσης ε, των ε, επενδύσεων όσον αφορά την ε, ανάπτυξη την οικονομική που πρέπει να επιτευχθεί. Τι να κάνουμε λοιπόν με αυτή την κατάσταση, να έχουμε εμπιστοσύνη στις αγορές, στις αγορές κεφαλαίων, όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι πολύ λίγα. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο διεθνές εμπόριο και στην απελευθέρωση των διεθνών συναλλαγών και θίγει ακριβώς αυτά τα ζητήματα ο εισηγητής που θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα δεν επέφεραν καμία αλλαγή και δεν επηρέασαν καθόλου την επίλυση των προβλημάτων χώρια από την αγορά εργασίας και την κατάσταση που υφίσταται στον δημόσιο τομέα σε όλους τους τομείς της οικονομίας όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα κτλ. Έχουμε σε αυτά όλα και με εμένα με ανησυχεί αυτό αυτή η πρόταση να συμπεριληφθεί εδώ πρέπει να συμπεριληφθεί μία ανησυχία για όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται σε σχέση με την αντιμετώπιση των ελλημάτων. Τι είναι αυτό το οποίο λέμε, ποιες κυρώσεις είναι αυτές και πώς θα επιβληθούν. Ήταν αυτή η θέση λοιπόν του Κοινοβουλίου. Αυτή θα είναι η οδός για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια συνένεση για αυτή την έκθεση. Εγώ θα λέγα ότι αυτή η πρόταση είναι σχεδόν προκλητική Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, για να προχωρήσουμε, εμείς φυσικά πόρο απέχουμε, πολύ μακριά απέχουμε από αυτή την έκθεση και φυσικά επιμένουμε και μένουμε στην ανάγκη μιας αναθεώρησης, ευφυούς αναθεώρησης αυτών των θεμάτων στρεφόμενοι στις ανάγκες αυτών των χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, που πρέπει να αντιστοιχίσουμε τις ανάγκες αυτών των χωρών σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να υπάρξει μια ανάκαμψη και να υπάρξει μια δυνατότητα να το σύνολο αυτών των χωρών να επωφεληθούν και όχι μόνο κάποιες χώρες από αυτές. Και εξάλλου αναφέρθηκε ότι ένα από τα κυριότερα προβλήματα αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυσικά θέτει εν αμφιβόλο την αξιοπιστία είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση σε σχέση με μια πολιτική και διαδικασία ολοκλήρωσης που δεν είναι καθόλου ουδέτερη και δεν είναι ισότιμη και ίση και ίδια για όλες τις χώρες. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων χωρών εις βάρος άλλων. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα. Ο κύριος Έικχουτ δεν είναι εδώ. Τότε ο κύριος Βάλλη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ διάβασα με πολύ προσοχή την έκθεση του Γκούναρ ε, σχετικά με αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ασχολούμαι με αυτό εδώ και τρία χρόνια και θέλω να σας πω ότι ε, Μία άποψη που είναι εκτεμέτρο αντίθετη με τη δική μας είναι αυτό που αναφέρεται για την ε, διακυβέρνηση. Ε, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και αυτά που ελέγχθησαν στην Ολομέλεια, τελευταία Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Άκουσα και τις ερωτήσεις του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως απαραίτητο να ε, προκαλέσουμε πραγματική ανάπτυξη χωρίς ε, πληθωρισμό τη στιγμή που έχουμε χαμηλές τιμές για τις πρώτες σύνδελες κάτι που δεν θα διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για άλλη μια φορά λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα στην νομισματική πολιτική, ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να αλλάξουμε πορεία. Αυτά που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση δυστυχώς ε, αφορούν μια προεκλογική εκστρατεία για αυτούς που ε, θα κατέβουν στις εκλογές στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Όμως εγώ πιστεύω ε, και ως ε, εκπρόσωπος της δικής μου της πολιτικής ομάδας ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετη αυτή η κατάσταση. Αντί να ζητάμε δημόσιες επενδύσεις για να δώσουμε κάποιο οξυγόνο στην Νότια Ευρώπη, ζητάμε να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες ε, και αυτό το ζητάει η Γερμανία που έχει την μεγαλύτερη ανισορροπία στη χώρα, στη ζώνη του ΕΜΒΡΟ. Και βεβαίως όλοι οι οικονομολόγοι με λίγη ευσυνειδησία, δεν αναφέρουμε σε ε, γενικούς ε, και σε ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί. Μιλάω σε αυτούς, ε, στο Στίγκλιτς και άλλους που έχουν κερδίσει βραβείο Νόμπελ και λένε ότι η Ευρωζώνη δεν μπορεί να σταθεί. Κατόπιν τούτου δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το σχέδιο το οποίο θα δημιουργήσει ανισορροπίες και ακόμα πιο σοβαρούς συμβιβασμούς που θα τιμωρήσουν τις ομάδες εκείνες οι οποίες θα στηρίξουν αυτό το πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής η οποία θα μας οδηγήσει στο να αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς κανόνες οι οποίοι όμως ε, κανόνες είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Κατόπιν τούτου πρέπει να αναθεωρηθούν αυτές οι απόψεις και οι δικέ μας οι τροπολογίες θα κατατεθούν προς αυτή την κατεύθυνση για να αποδείξουμε ότι η Ευρωζώνη και τεχνικά και πολιτικά ε, δεν μπορεί να στηριχθεί στο πλαίσιο μιας κρίσης. Οφείλουμε λοιπόν να ζητήσουμε κάτι το οποίο είναι, θεωρείται ιερό και άγιο, δηλαδή να γίνουν δημόσια επενδύσεις τουλάχιστον στις χώρες του Νότου, γιατί μόνο έτσι μπορεί να βελτιωθεί, να κατευναστεί λιγάκι η κατάσταση, αυτή η τραγική κατάσταση ε, στην οποία βρίσκονται οι νότιες χώρες. Μην ξεχνάτε, 60% των Ιταλών εχθές καταψήφισαν την κυβέρνηση η οποία ήθελε να εφαρμόσει αυτές τις ενωσιακές πολιτικές χωρίς να έχει κατά νου ε, το τι πραγματικά συμβαίνει. Η ε, μείωση των ε, μισθών. Αυτό ήταν μια συνέπεια, κάτι το οποίο το ζήτησαν οι γέρακες εκείνοι, τα γεράκια που βρίσκονται στο Συμβούλιο. Αν λοιπόν η Ευρώπη θέλει να επιβιώσει πρέπει να ξεπεράσει τέτοιου είδους δόγματα, αλλιώς οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτικές δυνάμεις που θα αναζητήσουν κάποιες άλλες λύσεις. Όσοι λοιπόν ε, προτείνουν κάτι τέτοια, πολύ σύντομα φοβάμαι δεν θα βρίσκονται στο ε, κοινοβούλιο μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάλλη. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητάει το λόγο. Εκτός... Α, ο κύριος Λάγκεν, παρακαλώ. Ποιος θα πάρει τώρα τον λόγο. Λάγκεν. Ζήτησα τον λόγο μετά από την τελευταία παρέμβαση, διότι ο συνάδελφος από την Ιταλία θεωρεί, επειδή έχει προβλήματα με μια, ένα δημοψήφισμα η Ιταλική κυβέρνηση, ο συνάδελφος ο οποίος ε, ε, καταθέτει μια έκθεση δεν θα πρέπει λέει να έχει έδρα στο μέλλον. Είναι μια ιδιαίτερη παρέμβαση αυτή, ιδιαίμορφου χαρακτήρα. Ζήτησα όμως τον λόγο για να πω κάτι άλλο σχετικά. ο απλός τύπος ότι το δημόσιο δηλαδή πρέπει λέει να επενδύει περισσότερα δεν είναι αποτελεσματική αυτή η διατύπωση. Πρέπει να έχουμε προγράμματα που θα έχουν όφελος για την ε, οικονομία και θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και μπορούμε σίγουρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πούμε ναι εντάξει τμήματα των ε, πολιτικών μας, των διαθωτικών πολιτικών ε, και με μέτρα υποδομής μπορούν να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα και η αναφορά σε σχέση με την θέση της Γερμανίας στην Ευρωζώνη δεν επαρκεί να πει κανείς τι όλα θα πρέπει να αναθεωρηθούν στα επιμέρους κράτη-μέλη. Μπορεί κανείς να πει ότι η Γερμανία έχει μάλλον υποεκτιμηθεί σε σχέση με την ισχύ της οικονομίας της. Πριν από 15 χρόνια αναφερόταν ότι η Γερμανία λέει θα γίνει ο ασθενής της Ευρώπης. Πράγμα στο οποίο ίσως οι Ιταλοί κατέληξαν ως ασθενείς της Ευρώπης σήμερα. Και ανελήφθη έγιναν μεταρρυθμίσεις στην Γερμανία σε σχέση και με την αναγκαιότητα να προσαρμοστεί η Γερμανία όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της. Δεν είναι μόνο για την Ευρωζώνη, είναι η ανταγωνιστικότητα έναντι και της, των ΙΠΑ και της Κίνας. Και δεν μπορεί κανείς απλά να λέει το κράτος να δίνει περισσότερα κονδύλια και έτσι θα επιλύονται όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό είμαι πεισμένος ότι χρειαζόμαστε μια νυφάλια αντικειμενική ανάλυση μια ε, καθαρή ματιά για τις επενδύσεις που χρειάζονται για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και κυρίως σε κάποια κράτη-μέλη χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις και σε αυτά μπορεί να ανήκει σίγουρα και η Γερμανία περαιτέρω. Ευχαριστώ. Η κυρία Πέρες. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποφαίνεται για την ετήσια αυτή έκθεση και ανησυχούν λιγάκι για τις προτάσεις του συγητή μας φέτος. Ίσως η αντίληψή του για την κατάσταση της Ευρωζώνης να είναι κάτι ξένο ως προς αυτόν. Διακόπτη κυρία Μπερές. Έλεγα λοιπόν ότι ο εισηγητής ίσως να μην ε, συνάδει με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωζώνη και αυτό είναι λάθος. Μα έχει τύχει και άλλη φορά να μην μπει τίποτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα ήθελα να μα συμβεί το ίδιο. Τώρα για τα όσα μα προτείνει συγκεκριμένα. Κάνει πίσω σε σχέση με πρόοδο που έχει επιτευχθεί, που έχει αποφέρει καρπούς τις προηγούμενες χρονιές, τις προηγούμενες διαδικασίες, για να εξετάσουμε όχι απαραίτητα την κάθε χώρα μέλος και κατά πόσο τηρεί το σύμφωνο σταθερότητας κατά γράμμα, αλλά και με μια προσέγγιση που είπε ότι είναι πιο χαλαρή αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ευφύης, έξυπνη και βοηθάει στη λειτουργία της Ευρωζώνης. Εισάγαμε μια ανάγνωση μιας συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης στην Ευρωζώνη. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική πρόοδος και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια ζητούσαμε να γίνει αυτό και κάθε βήμα προς τα πίσω για μένα θα ήταν σφάλμα. Ακούω από τον κύριο Χόκμαρ κάτι το οποίο λυπάμαι κύριε Σιγητά, αλλά μου φαίνεται πεπαλωμένο. Όταν λέτε ότι η νομισματική πολιτική έχει φτάσει στα όρια της, μα αν η νομισματική πολιτική έχει φτάσει στα όρια της, τότε θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο και εσείς προτείνετε απλώς και μόνο να είναι οι χώρες μέλη οι οποίες θα εφαρμόσουν πολιτικές ανταγωνιστικότητας όπως λέτε. Ναι, αλλά γνωρίζετε ότι αν οι χώρες δεν κάνουν τίποτα λεκτό από αυτό, τότε μπαίνουμε σε ένα σπιράλ υποτίμησης, εσωτερικής υποτίμησης μεταξύ χωρών μελών που δεν θα οδηγήσει πουθενά. Παρά μόνο θα μας βάλει πάλι σε κίνδυνο ύφεσης. Και κατά κάποιο τρόπο μια ερώτηση θέλω να κάνω στον εισηγητή. Γιατί έχουμε το σχέδιο Juncker και γιατί όλοι συμφωνούν και λένε ότι πρέπει να νεωθεί αυτό το σχέδιο Juncker, μάλλον γιατί νιώθουν ότι χρειάζονται επενδύσει στην Ευρωζώνη. Οπότε, πέρα από το σχέδιο Juncker, δεν νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους προσανατολισμούς που δίνει για την λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά πρώτον και δεύτερο κατά χώρα ότι θα έπρεπε να λάβει υπόψη αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάν. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση καθοριστική σημασίας κατά την άποψή μου. Δουλεύουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο βασίστηκε στην εμπειρία των γεγονότων της αρχής της δεκαετίας του 90. Δεν πιστεύει ο εισηγητής ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο κριτική προσέγγιση. Τα οικονομικά, κοινωνικά, χρηματοπιστωτικά κριτήρια της αρχής της δεκαετίας του 90 εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να ασκήσουμε κριτική στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για το κατά πόσον αυτά πράγματι βοηθούν στο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Πιστεύετε ότι έχουμε μια πραγματική εικόνα της, μια εικόνα της πραγματικότητας του που πρέπει να απαντήσουμε, το τι πρέπει να κάνουμε για να υπάρξουν επενδύσεις, να υπάρξουν θέσεις απασχόλησης. Πρόσφατα είχαμε τον διοικητή της ε, Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε για κυκλική μείωση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ, κυκλική μείωση των επενδύσεων, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών. Και είπε ότι δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτή η μείωση. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι θα έπρεπε ίσως και να συζητήσουμε τις μεθόδους ε, που χρησιμοποιούμε, ε, την προσέγγιση που προβάλλουμε. Βεβαίως, μην ξεχνάμε και την νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα στην οποία ζούμε, αλλά σε τελική ανάλυση υπάρχουν και ξεπερασμένες έννοιες όσον αφορά την πραγματικότητα. Τώρα ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας των 90. Η παγκοσμιοποίηση έχει προχωρήσει με ταχύτατο βήμα και οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτά που κάνουμε δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ε, ίσως ε, να προβάλλουμε ιδέες που έχουν σχέση με τα ολιγοπόλια σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά αυτό θέλουμε τελικά και αυτή είναι η τάση που επικρατεί όλο και περισσότερο. Ό,τι και να κάνουμε δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των πολιτών, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών ολιγοπολίων. Δεν πιστεύει λοιπόν η συγητής ότι έχει φτάσει πια η στιγμή να δούμε τα πράγματα με κριτικό μάτι, ε, τουλάχιστον για να αναζητήσουμε κάποια λύση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαν. Άλλος κανείς? Κανείς. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στον ε, εισηγητή μας για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ο κύριο Χοκμέρ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για τον προβληματισμό και για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να στραφώ στην κυρία Μπερές. Το σχέδιο Juncker υπάρχει γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς εδώ που να πιστεύει ότι μπορούμε να πετύχουμε και το επίπεδο επενδύσεων στην Ευρώπη δαπανώντας από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή από το δημόσιο τομέα. Χρειαζόμαστε ιδιωτικέ επενδύσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε σταθερότητα και χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη προοπτική χαμηλών επιτοκίων. Επιτρέψτε μου επίσης να επενθυμίσω τι έγινε. Όταν ήμασταν πολύ ελαστικοί με την ε, πολιτική μας τον προπολογισμό, τι έγινε στις διάφορες χώρες και έγινε στις περισσότερες χώρες μας όπου υψηλά ελλείμματα και το υψηλό επίπεδο ευελιξίας, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, είχαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η Γαλλία και η Γερμανία έμειναν απ' έξω. Ναι, δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, αλλά όπου αυξήθηκαν τα ελλείμματα, δεν βλέπαμε επενδύσεις. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Να δούμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Είχαμε 8 χώρες μέλη σε υπερβολικό έλλειμμα δεν οδήγησε αυτό σε επενδύσεις, σε ανάπτυξη. Οδήγησε σε μεγαλύτερα ελλείμματα και άνοιξε το δρόμο στη λιτότητα. Γιατί όταν δεν μπορείς να δανειστείς, δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις, τότε καταλήγεις σε δρακόντια μέτρα λιτότητας. Αυτό το οποίο χρειάζεται, αν θέλουμε να πετύχουμε συμφωνία, και ελπίζω ότι θα το πετύχουμε, με την πλειοψηφία τουλάχιστον εδώ, πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο δεν θα αντιμετωπίσουμε παρά μόνο αν βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, βελτιώσουμε την καινοτομία μας, τις επενδύσεις μας από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί γνωρίζουμε ότι στην παγκόσμια οικονομία υπάρχουν χρήματα, αλλά πρέπει να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Αν χάσουμε τον έλεγχο των ε, δημοσιονομικών μας, των δημοσίων οικονομικών, ε, τότε δείχνουμε ότι χάνουμε τον έλεγχο και γινόμαστε μία απειλή κατά της ε, αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν είμαστε απειλή απέναντι σε κανέναν άλλον. Με τα ελλείμματα που είχαμε δεν πετύχαμε να δώσουμε κίνητρα. Όπου αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα, επανήλθε η ανάπτυξη. Είχαμε ανάκαμψη της οικονομίας. Δεν πρέπει να συζητάμε μόνο το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά να συζητάμε και για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να ελπίσουμε ή να έχουμε σαν άλοθη, δεν κάνουμε δηλαδή ε, διαρθρωτικές αλλαγές ε, γιατί θα βοηθήσει η δημοσιονομική πολιτική. Όχι. Αυτό μόνο προβλήματα σε λιτότητα και κοινωνικής πολιτικής. Φυσικά πρέπει να δούμε και στις χώρες εκείνες που έχουν περιθώριο να χρησιμοποιήσουν δημοσιονομικά εργαλεία. Τι θα πούμε στις οικονομικές αγορές, ότι δεν θέλουμε πια σταθερότητα μέσω κανόνων. Πρώτα απ' όλα έχουμε νομοθεσία και έτσι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην νομοθεσία μας. Αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε καρποφόρα συζήτηση για το πώς θα διασφαλίσουμε ε, καθορισμό προπολογισμού ποιότητας, με διαρθρωτικές αλλαγές, με προσέλκυση επενδύσεων. Αλλά πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες που έχουμε. Γιατί αλλιώς υπονομεύουμε τη σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ που είστε ευγενεί, κυρία Μπέρε. Λέει ο κύριο Χόκμαρ σε παρέμβαση χωρί μικρόφωνο τη κυρία Μπέρε. Οι τελήματα δεν θα βοηθήσουν. Ε, ο πρόεδρο Μάτο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χόκμαρ. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω πριν ολοκληρώσουμε το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 14 στις 12 το μεσημέρι. 14 του μηνός στις 12 το μεσημέρι. Στις 12 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε τι τροπολογίε, θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ στις 6 Φεβρουαρίου και προβλέπεται να πάει το θέμα στην Ολομέλεια στις 13 Φεβρουαρίου. Εντάξει. Ωραία. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και το επόμενο προβλέπεται για τις 5, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 5 λεπτό και θα είμαστε και πάλι εδώ στις 5 ακριβώς.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 Good afternoon, dear colleagues. Σας απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να περάσουμε τώρα. Δεν βρίσκω το σφυράκι. Πού είναι? Okay. But um, I would like to welcome, please, colleagues, could you be silent, please? Thank you. Ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω την Έλκε Κόνιχ, πρόεδρο του ε, Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης ε, Single Resolution Board που ήρθε η κυρία Κόνιχ ε, με την παρουσίαση του, της ετήσιας έκθεσης κατά τον Ιούλιο. Τώρα έρχεται μετά τη δημοσίευση του προγράμματος εργασίας για το 2017 από πλευρά SRB. Και αυτή τη στιγμή γίνονται πολλά για το πρόγραμμα εργασιών του Single Resolution Board και έχουμε συνειδητοποιήσει πάρα πολύ το θέμα των ε, νομοθετικών μέτρων που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με διάφορα θέματα και για τον ε, συντονισμό μεταξύ αυτών. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Σας δίνω αμέσως τον λόγο λοιπόν ε, κυρία Έλκε Κένιχ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές με μεγάλη ικανοποίηση βρίσκομαι ενώπιον σας. Δεν πέρασε πάρα πολύς χρόνος από ό,τι φαίνεται από την τελευταία φορά, αλλά έχετε δίκιο. Τουλάχιστον είναι η τέταρτη επίσημη ακρόαση, ακροματική διαδικασία από τότε που το SRB ε, κατατίστηκε, συγκροτήθηκε. Περνάω μέσα στην ουσία του θέματος. 200 αναπτύσσουμε την οργάνωσή μας και 200 δημιουργούμε όλο και περισσότερο τις προϋποθέσεις ε, για το ταμείο αυτό, το FUND, για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά για να είμαστε ρεαλιστές πολλά πρέπει ακόμα να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να γίνουν του χρόνου και τα επόμενα χρόνια καλύτερα. Και θα στραφώ αμέσως στο θέμα το οποίο μας απασχολεί και είναι ε, του ενδιαφέροντος για ε, την απόψινή συνεδρίαση. Στρεφόμαστε προς το μέλλον ως ε, οργάνωση σε σχέση με την ε, ε, εξυγίανση και διευθέτηση και έρχομαι μετά από μια διευρυμένη εκτελεστική συνεδρίαση όπου συζητήσαμε αυτά τα θέματα σε σχέση με το 2016. Ολοκληρώνουμε αυτή τη στιγμή τον πρώτο γύρο υπό τις ευθύνε μας και ε, οικοδομούμε στο πολύ καλό έργο που έγινε από τις ε, εθνικές ε, αρχές Resolution Authorities κατά το παρελθόν. Κατά τα τέλη του έτους ελπίζουμε ότι 70 τέτοια προγράμματα και σχέδια θα έχουμε εγκρίνει και για 30 περαιτέρω μεταβατικά τέτοια προγράμματα, δηλαδή σε σχέση με τον πρώτο γύρο, όμως πιο εξειδικευμένα αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλύψει μεγάλο βαθμό των ε, υποχρεώσεών μας. Όμως αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ε, υλοποιήθηκε η εντολή και ολοκληρώθηκε. Ξεκινήσαμε και όπως ε, αναφέρθηκε είναι μια διαδικασία και όχι ένα τελικό προϊόν, μια ενρευστό διαδικασία υποεξέλιξη. Σε σχέση λοιπόν με τις ε, στρατηγικές αυτές και δημιουργώντας ε, ελάχιστες προϋποθέσεις και απαιτήσει για αυτές τις υποχρεώσεις θα απαιτήσει χρόνο συνολικά. Το 2017 θέλουμε και πρέπει να έχει επιτευχθεί πρόοδος για την στρατηγική μας. Πρέπει να είμαστε πιο εξειδικευμένοι, πιο α, καταλεπτός εργαζόμενοι στα εργαλεία και στους στόχους μας και να αντιμετωπίζουμε τα προσκόμματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Άλλο είναι το ότι πρέπει να λέει κανείς ότι μπορούμε να έχουμε μια ανοιχτή διαδικασία bail-in για την ε, διάσωση και είναι ένα άλλο πράγμα να λέει κανείς εδώ υπάρχει ένα πρόσκομα, ένα εμπόδιο και πρέπει να το υπερβούμε. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν προγράμματα και σχέδια για το σύνολο των αρμοδιοτήτων μας και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα για την ολοκλήρωση της στρατηγικής μας. Και σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε internal benchmarking, τις βέλτιστες προδιαγραφές, ώστε όλες, όλα τα προγράμματα και τα σχέδια να αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη συνέπεια. Όλα αυτά τι σημαίνουν την υιοθέτηση των κατοφλίων και προδιαγραφών. Αυτό είναι κέρια σημασία για τον ρόλο μας ε, όσον αφορά τον, ε, το όργανο ε, εξυγίανσης στον τομέα μας. Είμαστε το όργανο για να επιτευχθεί αυτή η εξυγίανση σε σχέση με τραπεζικά ιδρύματα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει δυνατότητα αφομοίωσης ε, των κραδασμών ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις ε, ε, κέρυες οικονομικές λειτουργίες χωρίς να υπάρχει ζημία στα χρήματα των φορολογουμένων. Δεν υπάρχει ένα μέτρο το οποίο ισοπεδωτικά να μπορεί να υιοθετηθεί για όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένη η δράση μας ανάλογα με τις ανάγκες επιτρέψτε μου να τονίσω ε, το ρόλο του ως αρχή να μπορούμε με επαρκή διακριτική ευχέρεια να κρίνουμε το τι πρέπει να γίνεται και τώρα ακολουθεί ε, μια πρόταση που αυξάνει την πίεση. Δηλαδή ένα 8% σε σχέση με τις συλλογικές ε, αυτές υποχρεώσεις όμως αναπερίπτωση θα πρέπει να εξετάσουμε το τι θα απαιτείται για τις μεγαλύτερες τράπεζες. Να θυμόσαστε ότι αυτό το 8% σε εμπόδιο ή ως κατόφλι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται στο Ταμείο και κανείς από εμά δεν θέλει όταν ξεκινά μια τέτοια διαδικασία να αναγνωρίσει ότι δεν θα υπάρχουν επαρκώς ρευστά ε, και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε από τη δειγματοληψία τραπεζών που εξετάσαμε μέχρι τούδε, εξετάσαμε σε βάθος ε, και είδαμε σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους και τις δομές τους το τι συμβαίνει και καθορισμό ελάχιστων προαπαιτήσεων σε σχέση με τις ε, κατεντολήν πράξεις, κατεξουσιοδότηση πράξεις και με βάση όλα αυτά κάναμε μια πρώτη αξιολόγηση. Και όλα αυτά θα πρέπει βέβαια κουμγκράνο άλλη να ε, εξετάζονται με ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Ε, το 8% θα ήταν ένας δεσμευτικός όρος περιοριστικός στις περισσότερες περιπτώσεις το 8% είναι κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο το οποίο θα απαιτεί το με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις Το 2017 πρέπει να συνεχίσουμε με το έμρο, δηλαδή από μια ομάδα θα πρέπει να περάσουμε στις επιμέρους, ε, στους επιμέρους ε, φορείς υπό την ε, ε, ένταξη αυτή και θα πρέπει να δούμε πώς αυτό θα εντάσσεται μέσα στους τραπεζικούς κανονισμούς ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει με το βέλτιστο τρόπο. Για ένα πιο σύντομο σχόλιο όσον αφορά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή, δημιουργεί μια σαφήνεια σε σχέση με το μέλλον όπως στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πώς θα πρέπει λοιπόν σε σχέση με αυτό να διευθετείται με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και εξετάζοντας αυτά είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να ανατρέπει το έμρο, ούτε θα πρέπει να το ε, καθιστά παροχημένο ή να θεωρήσουμε ότι μπορεί να είναι ανεδαφικό. Αυτό τουλάχιστον με την πρώτη μας ανάγνωση. Η πρόταση υπογραμμίζει το ότι πρέπει οι τράπεζες ε, να μπορούν να εξηγιανθούν αποτελεσματικά θα το εξετάσουμε αυτό διαμακρόν. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Η, ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερα όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα και τις, ε, γιατί υπάρχει και μια δεύτερη ε, δομή που είναι σημαντική σε σχέση με την Ευρώπη και βλέπουμε το πώς πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία υλοποίησης και συνδέω αυτό με το πρώτο σχόλιο, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αναγκαία ελαστικότητα, σε σχέση με τις αρχές εξυγίανσης, ώστε να έχουμε ένα αποτελεσματικό μέσο στα χέρια μας για να μπορέσουμε να καταστήσουμε υγιείς τις τράπεζες. Σε σχέση λοιπόν με τις προτάσεις αυτές από πλευράς συνομοθετών και του Ευρωκοινοβουλίου δηλαδή το σημερινό πλαίσιο υφίσταται και μας δεσμεύει και ως τελευταία τοποθέτηση έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε συγκεκριμένες αγορές ή από συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα και λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις προκλήσεις. Πρέπει να υπάρχει μια πιο ισχυρή, ένα πιο ισχυρό καθεστώς και πιο αξιόπιστο καθεστώς εξυγίανσης σε σχέση με τις τράπεζες από ότι το σημερινό τούτων λεχθέντων έχουμε ισχυρές τράπεζες. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν για ένα καθεστώς ισχυρών τραπεζών, υγιών τραπεζών Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε ετοιμότητα για να προβούμε σε αυτές τις εξηγιαντικές ε, δράσεις. Πρέπει να δούμε και με τους εταίρους μας ε, SSM, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ υφίσταται θετική συνεργασία, αλλά πρέπει σε καθημερινή βάση να συνεργαζόμαστε για να έχουμε μια αποτελεσματική διαδικασία πετύχαμε και μπορείτε να το δείτε αυτό αντικειμενικά ότι υπάρχει και ένα εγχείρημα στο οποίο αποδιόμεθα για την διαχείριση κρίσεων τράπεζες εκτός της ζώνης ευρώ ή εκτός Ευρώπης, ποια θα ήταν η αντίδραση και οι επιπτώσεις ήταν ένα, είναι ένα πολύ θετικό input και πρέπει να δούμε σε σχέση με τις αρχές τρίτων κρατών ε, διότι δεν σταματούν οι δραστηριότητες στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Και είναι ο τρίτος πυλώνας της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης που βρίσκεται υπό οικοδόμηση και υπό εξέλιξη. Χρειάζεται μια λειτουργία αντιμετώπισης προβλημάτων ώστε να λειτουργεί το σύστημα εγγυήσεων και να είναι κάτι παραπάνω από απλές δεσμεύσεις. Να είμαστε αποτελεσματικοί ε, στο σύστημα φερεγγιότητας ώστε να μπορέσουμε να ακολουθούμε τα πραγματικά αναγκαία μέτρα για να είμαστε αποτελεσματικοί. Και σημειώσαμε ότι ξεκίνησε το έργο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την statutory subordination δηλαδή την καταστατική ένταξη ή ε, ιεραρχία, ώστε να μπορούν να επιληθούν ζητήματα στο αντίστοιχο επίπεδο αρμοδιότητας και ιεραρχικής δικαιοδοσίας. Ένα τελευταίο σχόλιο το οποίο δεν είναι τόσο ε, στην δική μας ε, ε, εξουσία, είναι η εξυγίανση όπου συνεργαζόμαστε ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με την ύπαρξη σαφών κανόνων και κανονισμών για την εξυγίανση. Και το τελευταίο μου σχόλιο θα είναι για το Ταμείο. Έχουμε 10,8 δις τα οποία συνελέγησαν σε σχέση με τις μεταφορές για το 2015 έχουν όλες οι μεταφορές ολοκληρωθεί για το 2016 από τις εισφορές που συνελέγησαν και που βρίσκονται στο ταμείο μας και για τη διαδικασία του 2017 που μόλις ξεκίνησε ήδη όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ σύνθετη περίπλοκη διαδικασία και εργαζόμαστε σκληρά ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ε, διαφάνεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν σε ετοιμότητα να ξεκινήσουμε όταν θα είναι έτοιμα και τα κράτη-μέλη. Ολοκληρώνω εδώ γνωρίζοντας ότι έχω υπερβεί το χρόνο μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμεί σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχατε πάρα πολλά θέματα που έπρεπε και θέλατε να θίξετε. Απαραίτητο θα έλεγα μάλιστα. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις ε, ερωταπαντήσεις. Αλλά πρώτα ε, πρέπει να σας ε, ενημερώσω ότι αυτή την Πέμπτη στις 8.30 θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με τη ΛΥΜΠΕ για να προτείνουμε ε, την ψηφοφορία, της ψήφου σχετικά με τις ε, κατεξιότητες πράξεις ε, blacklist. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Κιονίχ που ήρθε. Δεν τα έχω μετρήσει ακριβώς πόσες φορές ε, έχετε έρθει, αλλά ξέρω ότι ε, με μεγάλη χαρά έρχεστε. Και ευχαριστούμε και για την ετήσια έκθεση. Σχετικά με το πακέτο μείωση κινδύνου, μιλήσατε για το TELAC και το ΑΜΡΕΛ, αλλά ίσω μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε και τι αλλαγέ του άρθρου 55 στην EBRD το πακέτο που περιλαμβάνει τα MRL και το TLAC, ε, τι ακριβώς πιστεύετε από αυτού. Πιστεύετε ότι αρκούν αυτά και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την προσαρμογή του DGS μέσα στο πλαίσιο των MREL. Μπορείτε λιγάκι να διευκρινίσετε την ε, προσαρμογή των DGS όταν θα καθορίζονται τα MREL. Ε, ξέρουμε πώς αυτά είναι στη θεωρία, αλλά μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς αυτά θα λειτουργήσουν στην πράξη. Και αν μετά ε, το DGS γίνει πιστοτής σε μια διαδικασία. Μήπως μπορείτε να μας διευκρινίσετε τη διαδικασία. Ξέρετε ότι δουλεύω σκληρά για το σύστημα EDIS και δουλεύουμε στο πώς θα λειτουργεί το σύστημα και μπορούν να επιστρέψουν κονδύλια στο σύστημα. Ίσως αυτό μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε. Και κάτι πιο εύκολο. Μετά το δημοψήφισμα στην Ιταλία, πώς ακριβώς αξιολογείται τον κίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ξεκινώντας από την αρχή. Το πακέτο μείωσης κινδύνου, άρθρο 55. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, πρέπει να πω ότι εξακολουθούμε να αναλύουμε το πακέτο. Όσον αφορά το άρθρο 55, εμείς ανέκαθεν συμφωνούσαμε ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το άρθρο 55 ε, στη διατύπωσή του δεν έχει ε, καθόλου αποκλεισμού, είναι πάρα πολύ γενικό και τώρα πρέπει να το αναθεωρήσουμε ε, για να υπάρξει αναγνώριση σε ευρύτερη κλίμακα θα πρέπει να υπάρξει κάποια προσαρμογή subordination. Ε, όλοι γνωρίζουν, όσοι με έχουν ακούσει, έχουν ακούσει να λέω ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή λύση, μια λύση που θα ε, λύσει γρήγορα το πρόβλημα. Τώρα το πρόβλημα που έχει τεθεί μοιάζει λιγάκι με την γαλλική νομική πρόταση. Άλλες προτάσεις παραμένουν ενισχύ, αλλά είναι μια πρόταση που χρειάζεται λίγο χρόνο έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα του ενδιάμεσου. Εγώ λοιπόν ε, θεωρώ ότι μια αρχή εξυγίανσης ποτέ δεν είναι ικανοποιημένη και αν τελικά βρούμε μια καλύτερη λύση ακόμα καλύτερα. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. προσαρμογή του DGS ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη εδώ γιατί αλλιώς θα πανικοβληθεί η ε, ομάδα μου, οι συνεργάτες μου, να σας απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, γραπτά ε, σε αυτό το θέμα, γιατί μόλις αρχίσαμε να το εξετάζουμε το θέμα, θα σας δώσουμε μια γραπτή απάντηση πριν σας πω ανοησίες. Και τέλος, ε, σχετικά με την τελευταία σας ερώτηση, κοιτάξτε το δημοψήφισμα, ήταν πολιτικό, οι αγορές είναι ήρεμες σήμερα, και εγώ δεν θεωρώ ότι το δημοψήφισμα έχει άμεση σχέση με τις ε, καθημερινές μας διεργασίες. Πολ Τάγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ την κυρία Κένινγκ. Δύο σημεία πολλά θα μπορούσα να ρωτήσω, αλλά θα επανέλθω στο έντις. Και την αμοιβεοποίηση που λέγαμε ότι δεν επηρεάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως αυτή η ανάλυση επιπτώσεων σημαίνει ότι υπάρχει αμοιβοποίηση των ταμείων. Εσείς λοιπόν πώς βλέπετε τη δυνατότητα μεικτών ε, ταμείων στο στάδιο 3, εθνικών και ευρωπαϊκών δηλαδή. Θα ήθελα τη συμβουλή σας και τα σχόλιά σας από αυτού. Το δεύτερο. Ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης αναφερόταν σε μεταφορές από εθνικά ελεκτικά συνέδρια στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Όμως η αποτελεσματικότητα και οι δυνατότητες απαλλαγής δεν φτάνουν. Και έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου λέει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εσεί ότι υπάρχει ένα κενό δηλαδή ελέγχου. Εσεί πώ το αξιολογείτε αυτό στον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2. Δεν είναι εύκολε οι σα σας σήμερα, λέει κύριε Κένε, για το TGS. Διάβασα την έκθεση του συγητή. Δεν πρόκειται για ένα θέμα όπου εμείς ως SRB, ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, το έχουμε σαν δικό μας θέμα. Υπάρχει η αμοιβεποίηση για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι για να βγούμε από τις συμφωνίες διευκόλυνσης δανείων μέχρι το επόμενο στάδιο. Αυτό θεωρούμε δεδομένο. Εγώ διάβασα την μελέτη επιπτώσεων που μιλάει για πλήρη αμεβεοποίηση, αλλά ήδη είμαστε πολύ κοντά. Και αυτό σημειώνω εγώ, ότι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά στο πρόγραμμα εργασίας σας, εσείς συνεισφέρετε. Πώς συνεισφέρετε χωρίς να μπορείτε να εκφέρετε γνώμη. Η γνώμη μου είναι ότι θέλω ένα λογικό τρόπο για να περάσουμε από πλήρως εθνικό επίπεδο, γιατί πάντα συζητούσαμε και λέγαμε ότι το Paybox είναι μία λειτουργία, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικά μέτρα. Η μεταφορά λοιπόν των καταθέσεων σε ένα άλλο όργανο είναι ένα μήνυμα έχοντας πάρει μαθήματα από κάποιους μη Ευρωπαίους συναδέρφους με πολύ περιορισμένες μεν λύσεις, αλλά πιο αποτελεσματικές από ό,τι φαίνεται. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα που οικοδομούμε βήμα-βήμα. Αλλά σημειώνω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτού. Και το άλλο θέμα που αναφέρατε, επίσης σημείωσε εδώ, για το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο και την έκθεσή του. Υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο SSM που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η ΜΟΝ που είμαστε υπηρεσία εδώ στις Βρυξέλλες. Και εμεί συζητάμε με το ελεγκτικό συνέδριο γιατί και εκείνοι κάνουν έλεγχο πάνω στο SRB, το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγένσης διότι αξιολογούν τα δεδομένα των ε, θεσμών. Έχουν το δικαίωμα εφόσον είναι Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Ελπίζω να απάντησα τουλάχιστον στη δεύτερη ερώτησή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. ECR δεν βλέπω. Η Σιλβιγκουλάρ. Καλή σας θα διατυπώσω την ερώτηση στα αγγλικά. Στο τελευταίο πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσφατα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν European Holding Companies. Θεωρείται χρήσιμη αυτή την πρόταση. Πώς αντιδράτε. Πώς θα έπρεπε να αντιδράσουμε ως νομοθέτες επ' αυτού για να σας βοηθήσουμε εμείς εσάς και όχι να δημιουργήσουμε προβλήματα. Ευχαριστώ. Ε, Πρώτα απ' όλα Καλό σας απόγευμα στα γερμανικά αντάπαντα. Και πάλι με τον όρο και προϋπόθεση ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης όλων αυτών. Όμως ουσιαστικά η ιδέα ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ένα συλλογικό σημείο εισαγωγής στον χώρο ευρώ έχει κάθε νόημα από πλευράς λειτουργίας. Σας δίνει μία προοπτική, σας δίνει τη δομή και σας λέει εδώ μπορείτε να δράσετε. Διαφορετικά θα είχαμε μία μονάδα εδώ, μία αλλού και θα ήταν μικρών διαστάσεων για να ε, τύχουν της προσοχής μας ε, ενώ ε, συνενούμενα θα έπρεπε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. Δεν έχω κάποια ετοιμικομένη ραμμένη απάντηση, πρέπει να την δούμε σε βάθος και μετά να τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Καλησπέρα σας, ε, Εμάση. Είπατε ότι πρόσφατα συναντηθήκαμε και έχω και εγώ αυτή την εντύπωση. Ε, συγγνώμη αν κάτι έχει ερωτηθεί, ε, τουλάχιστον μπορεί ίσως να έχει ε, διαφύγει απάντηση είσαστε σε θέση να μας δώσετε τις ε, εισφορές ε, των διαφορετικών τραπεζικών ε, ιδρυμάτων σε σχέση με τις διαστάσεις τους, σε σχέση με το ενιαίο σύστημα επίλυσης προβλημάτων. Θα μπορούσατε να μας τα διαθέσετε αυτά και δεύτερον για την ολοκλήρωση της Βασιλείας Τρία συμφωνίας. Θα συμφωνούσατε σε σχέση με τους κινδύνους modeling ότι υφίστανται ακόμα και πώς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να επιληθεί το πρόβλημα αυτό σε σχέση με τις ανησυχίες ότι η Βασιλεία 3 ή η Βασιλεία 4 θα μπορούσε να δημιουργήσει μειονεκτική θέση για τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα και ε, ε, επειδή δόθηκε κάποιο κίνητρο γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποια δεν ε, υπάρχει τοποθέτηση για την Ιταλία τουλάχιστον γίνεται η προσπάθεια αν θέλετε να συστήσετε κάτι στις Ιταλικές αρχές τι θα συνιστούσατε μια κεφαλαιοποίηση σε σχέση με την ε, τράπεζα Μόντε ε, τη Σιένα ή θα θέλατε να εξηγιανθεί ευθύ εξ αρχής. Να ξεκινήσω με την απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Δεν είμαι βέβαια ότι δώσαμε οποιασδήποτε λεπτομέρειες για τους τύπους ή τον τύπο τραπεζών. Έχουμε όμως αρκετές πληροφορίες ε, στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας και μπορώ να απλουστεύσω τα πράγματα, να σας αποστείλουμε αυτά τα στοιχεία στην ΕΚΟΝ με μια ε, κατηγοριοποίηση σε σχέση με τους ε, ε, τύπους κινδύνων και σε σχέση με τις ε, χώρες εκάστοτε. Θα πρέπει να ε, απόσχουμε από το να ε, ταυτοποιούνται άμεσα με βάση αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες οι οποίες ε, βρίσκονται πίσω από αυτά τα στοιχεία. Αν όμως σε σχέση με τις συστάσεις αυτές θέλετε κάποια στοιχεία θα σας τα διαθέσουμε μέσω ιστοσελίδας. Βασιλεία 3 ή Βασιλεία 4 όπως και αν το αποκαλέσετε θα ήθελα να απόσχω από σχόλια, διότι αυτό είναι δουλειά των εποπτικών αρχών. Όμως συμφωνώ παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα εσωτερικά πρότυπα και οι δομές και εδώ θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι το modeling δεν θα μπορούσε να έχει ε, κάποια να θεωρηθεί ως αυτός σκοπός. Από την άλλη πλευρά όμως δεν πρέπει τα ωφέλη να τα απεμπολούμε από μια θετική δράση και σε σχέση με ένα πρότυπο όπου δίνονται ίσως κίνητρα στις πιο επικίνδυνες, στις πιο ε, βεβαρημένες λόγω κινδύνων συναλλαγών. Ε, έχω λοιπόν την εμπιστοσύνη ότι με βάση τις γνώσεις τους ε, οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και τον Ιανουάριο να υποβάλουν, θα υποβάλουν μια τελική πρόταση. Και για την Ιταλία θα έλεγα κάτι το οποίο ίσως δεν θα σας εκπλήξει. Πάντα έλπιζα ότι οι τράπεζες θα έβρισκαν ιδιωτικές δυνατότητες λύσεων και εύχομαι κάθε επιτυχία σε τέτοιου είδους ιδιωτικές επιλύσεις προβλημάτων εναντί άλλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Σας ευχαριστώ. Σβεν Γκίγκολτ, παρακαλώ. Μάλιστα, καλό σας απόγευμα κυρία Κένιχε. αλλά θα συνεχίσω κι εγώ στα αγγλικά και όχι στα γερμανικά. Πρώτον, επειδή είναι η συνήθις ερώτηση προς εμάς. Μου είχατε υποσχεθεί πριν από καιρό έναν κατάλογο εμποδίων και προσκομμάτων στο εθνικό δίκαιο και ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με το έργο σας. Πότε θα μας υποβάλλετε αυτόν τον κατάλογο και πίνακα. Προτού ερωτήσω οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να απαντήσετε επ' αυτού συγκεκριμένα παρακαλώ με μια ημερομηνία. Να σας δώσω μια ημερομηνία σε σχέση με αυτό το θέμα δεν ε, θα ήταν ε, δυνατόν. Εργαζόμαστε ακόμα και ελπίζουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτόν τον κατάλογο για τα πρώτα προγράμματα εξυγίασης. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα εμπόδια τα οποία, τα οποία υφίστανται, όχι εμπόδια, όχι προσκόμματα, αλλά τομεί που πρέπει να εξεταστούν για να γίνουν τα πράγματα πιο λειτουργικά, είναι πολυσχηδείς αυτοί οι τομεί και πολυάριθμοι. Γι' αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμο αυτό ο κατάλογο. Μέχρι το καλοκαίρι επιτρέψτε μου να ευελπιστήσω ότι θα είναι έτοιμο ο κατάλογο. Αλλά είναι το καλύτερο που μπορώ να σα πω. Μπορώ να σα αποστείλω ένα μακρότατο κατάλογο για το ποια θα είναι τα θέματα για το 2017 που θα πρέπει να εξεταστούν και που θα πρέπει να καταστούν λειτουργικά με βάση τα ε, εξειδικευμένα στοιχεία. Και πάλι μπορώ να σας δώσω ένα εύκολο επιχείρημα ως απάντηση. Όταν υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθεσίας ε, ε, που ή δημιουργεί προβλήματα ή προκαλεί προσκόμματα η κατάσταση δεν επιλύεται. Σας υπόσχομαι ίσως την άνοιξη να σας υποβάλω ένα τέτοιο κατάλογο, όχι πλήρη κατάλογο αλλά τα πρώτα θέματα. Λοιπόν την άνοιξη θα μας δώσετε ένα πρώτο κατάλογο, πλήρη κατάλογο όμως μέχρι το καλοκαίρι. Τα συνοψίζω καλά πρώτος κατάλογος την Άνοιξη και ένας πιο επεκτα... ε, εκτεταμένος κατάλογος μέχρι το καλοκαίρι αναμένοντας ότι θα πρέπει τα προγράμματά μας να συνεχιστούν και να εξειδικευθούν Giggled. Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα αυτά θα έχουμε ένα αστείο βίντεο με αυτό το γύρο ερωτήσεων απαντήσεων ε, κατά τη χρονική αυτή διάρκεια των μηνών που περνούν και από πλευρά συναδέλφου που υπήρξε θύμα ενός τέτοιου βίντεο για την χρηματοδότηση Finance Watch. Πέραν αυτών όμως, πέραν αυτών θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δική μου εντύπωση, σε σχέση με αυτό, με αυτό τον κατάλογο από την Επιτροπή είναι ότι σας ε, ε, μειώνει τις δυνατότητες δράσης σας. Πώς ε, θεωρείτε ότι μπορούν ε, σε σχέση με θέματα τρίτων χωρών ε, να μπορέσετε να δράσετε πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα μέση που θα έχετε. Και με, για το κύλακ σε 6,75% αν μια τράπεζα έχει στον ισολογισμό της 18,5% του συνολικού αυτού απολογισμού θα βρίσκεται κάτω από το 8% έμρολ το οποίο πάντα προαναγγέλατε. Πώς το αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής από πλευράς της για να σας υποστηρίξουμε στο έργο σας είσαστε φιέστατος στο να επισημαίνετε αυτό το ένα σημείο το οποίο πολύ σύντομα προσπάθησα να καλύψω στην παρουσίασή μου. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τύχουν προσεκτικής αντιμετώπισης. Το ότι πιστά μετέφρασε το, τυπολόγιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά σε ένα ελάχιστο επίπεδο στον πρώτο πυλώνα και μετά προσέθεσε και ένα δεύτερο πυλώνα. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με αυτό. Όταν υπάρχει θέμα διακριτικής ευχέρειας από μια αρχή θα πρέπει να δικαιολογείται γιατί πρέπει ένα επίπεδο να είναι υψηλότερο ε, μιας ε, πρότασης που έχει τεθεί όπως για το Emerald που δεν είναι το ότι θα πρέπει κάποιος να ε, αναρριχηθεί σε μια κορυφή σε σχέση με το, με το δεύτερο πυλώνα τώρα που συνοδεύει τον πρώτο πάντα σε σχέση με την ευθυγράμμιση μιας πολιτικής για την εξυγίανση. Όταν έχουμε τον έναν πυλώνα για ε, DSIPs και δημιουργείται ένας δεύτερος πυλώνας ε, για τις υπόλοιπες υποθέσεις, πρέπει να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα θεωρηθεί ότι αφορά μόνο τις πολύ μεγάλες τράπεζες, το Emerald για τον πρώτο πυλώνα και για τις όλες μικρότερες τράπεζες θα ισχύει ο δεύτερος πυλώνας. Δεν είναι κάτι τέτοιο η πρόθεση, όμως η διατύπωση πρέπει να είναι σαφής και εύληπτη ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα Emerald αντίστοιχο με εκείνο το οποίο είχε τεθεί στην πρώτη προσέγγιση μας. Είναι κάτι που πρέπει λοιπόν να τελούμε ενεγρηγόρση επ' αυτού και για την ε, ε, ένταξη σε ένα ιεραρχικό πλαίσιο, subordination, ε, πρέπει να είμαστε και εδώ προσεκτικοί. Πάλι πρέπει να εξετάζονται οι επιμέρους ε, καταστάσεις και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ένταξη ιεραρχική των υπολείπων είναι αυτό το οποίο είπαμε. Πρέπει να δικαιολογούνται οι αποφάσεις ε, με αντικειμενικά κριτήρια. Και πάλι όμως θα έλεγα ότι να μην δημιουργηθούν επιπρόσθετα προσκόμματα και εμπόδια, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιθυμεί η Επιτροπή με την προσέγγιση της. Ευχαριστώ. Eh, Κοζάνη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των Ιταλικών ε, τραπεζών. Εσείς ε, απαντήσατε και ο κύριο Ντεμάζη είπε επίση ότι ελπίζει ότι θα υπάρξει μια λύση από την αγορά. Όμως ε, η ελπίδα δεν είναι πάντα η καλύτερη στρατηγική γιατί υπάρχουν και άλλες καλύτερες λύσεις ε, καλύτερη από την ε, ελπίδα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι αναβάλλεται η ανακεφαλοποίηση της Monte Τεϊπάσκη και εκεί προστίθεται και ένα πακέτο των μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ε, σε τιμές όμως που δεν ανταποκρίνονται στην αγορά. Στην περίπτωση όπου το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να στηρίξει με δημόσια κονδύλια μία τράπεζα, τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που η SRB αποφάσιζε να τοποθετηθεί σχετικά με αυτή την δημόσια χρηματοδότηση και στην περίπτωση που η Ιταλία θα αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει ένα ε, ιδιωτικό φορέα για να ανακεφαλαιοποιήσει μια τράπεζα. Ε, στην περίπτωση αυτή τι θα γίνει, θα ε, προέκυπτε αυτόματα το BRLD. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω και έχει πάντα σχέση με την Ιταλία είναι ένα καθοριστική σημασία θέμα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύστησε σε πολλέ Ιταλικέ τράπεζε να ξεφορτωθούν ε, κάποια ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η τιμή που θα πολιθούν αυτά τα πακέτα, δηλαδή ζήτηση και προσφορά. Η Monte dei Paschi, όπως λέτε και εσείς, ε, έχει το 37% αυτών των ε, μη εξημεριτούμενων ε, δανείων. Τον ε, Δεκέμβρη του 2015 είχε προταθεί μια τιμή περίπου στο 17,5% και μετά ανέβηκε αυτό στο 21%. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν και με βάση τα δικά σας τα προγράμματα εξυγίανσης για την Ιταλία, ποιο θα μπορούσε να είναι, ποια θα μπορούσε να είναι μια ικανοποιητική τιμή των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα απολυθούν, λαμβάνοντας ε, υπόψη ότι υπάρχει και πίεση ε, ουσιαστική αλλά και χρονική εις βάρος των Ιταλικών τραπεζών. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω την κατάσταση οποιασδήποτε τράπεζας. Αν δούμε λιγάκι την κατάσταση, όχι μόνο στην Ιταλία, υπάρχει ισχύει ένα πράγμα. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τους κανόνες. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχουν πάντα λύσεις ε, στον ιδιωτικό τομέα. Αν όχι, τότε η BERD και ο δικός μας ο προβλέπει εναλλακτικέ λύσεις. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι προληπτική ανακεφαλαιοποίηση, σε άλλες πάλι περιπτώσεις αν χρησιμοποιηθούν δημόσια κονδύλια, αν δεν είναι δηλαδή προληπτική ανακεφαλαιοποίηση, στην άλλη περίπτωση η τράπεζα είναι υποεξυγίανση. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει και το στοιχείο του επιμερισμού βαρών. Σε αυτή τη λύση δηλαδή. Και εμείς παρακολουθούμε στενά τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, και τις ανακοινώσεις της τράπεζας για το ότι όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στην Ιταλία οι τράπεζες οι οποίες έχουν εγγράψει στα βιβλία τους μεγάλα ποσά για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οφείλουν οι τράπεζες αυτές να τα μειώσουν. Ε, αυτή η μείωση δεν θα γίνει δωρεάν. Αν γίνονταν δωρεάν δεν θα υπήρχε και πρόβλημα αλλά σας λέω υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Για να είμαστε ειλικρινεί στα προγράμματά μας της εξυγίανσης, αυτό πάντα είναι ένα θέμα. Εμείς ε, προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας με βάση τις ανάγκες και τώρα πρέπει να σας πω δεν υπάρχει μία τιμή για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που να ισχύει ε, για όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν μάλιστα και πολλές διαφορετικές απόψεις ε, για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Σας λέω, δεν μπορεί να υπάρξει μια τιμή για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που να βολεύει σε όλες τις περιπτώσεις. Πάντως, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρξει εξυγίανση, λύση και όχι κάτι το οποίο να πρέπει κανείς ε, σύντομα να αναπροσαρμόσει και πάλι και πάλι. Ελπίζω λοιπόν ε, στην περίπτωση αυτή να επιλεχθεί από την αρχή η καλή λύση. Για να είμαστε όμως και λιγάκι πιο θετικοί, ε, κοιτάξτε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι λύσεις του ιδιωτικού τομέα είναι η καλύτερη λύση. Μπερνά Μονό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δύο θέματα. Πρώτον, το καθήκον του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης σίγουρα δεν είναι απλό, διότι υπάρχουν πολλές μεγάλες τράπεζες και υπάρχουν λίγοι υπάλληλοι οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα διασυνοριακά, με το τραπεζικό καθεστώς και τους πιστωτές. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα σε τράπεζες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα φέρετε σε πέρα στην αποστολή σας. Η εξυγίανση γίνεται στο φυσικό πλαίσιο που ανήκουν, δηλαδή στη χώρα μέλος. Εσείς πώς θα το κάνετε αυτό, για να μην πούμε για την Ιταλία, μετά το όχι κινδυνεύει να υπάρξει ε, πρόβλημα με τα πέντε δις που είναι τα κεφάλαια της ε, τράπεζας Μοτιντιπάτσι. Πώς θα βλέπετε εσείς τα πράγματα αυτά, θα πάρει την τράπεζα το κράτος, θα υπάρξει ε, μετάδοση σε άλλες τράπεζες και θα υπάρξει bail-in όπως προβλέπει η BBRD που θα ζητήσει από πιστωτές, δηλαδή από τους ε, Ιταλούς αποταμιευτές. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς την κατάσταση αυτή και πώς θα βλέπετε την εκλογική διαδικασία στην Ιταλία στην περίπτωση που αποφασιστεί το bail Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι θέλετε να με βάλετε να συζητήσω τις λύσεις για την Ιταλία. Θα προσπαθήσω ένα πράγμα να αποσαφηνίσω. Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο νέο Συμβούλιο Εξυγίανσης όταν πρόκειται για διασυνοριακές υποθέσεις. Και όταν λέω διασυνοριακές εννοώ μεταξύ ευρωπαϊκών ε, χωρών και μη ευρωπαϊκών χωρών. Εδώ εξακολουθούμε να δουλεύουμε με τους συναδέρφους μας, ώστε η εξυγίανση να αποτελεί λύση σε ένα θέμα. Άρα παραμένουμε μαζί, συνεργαζόμαστε και όχι το αντίθετο. Τώρα, αν πάμε πίσω στην περίπτωση που αναφέρατε για τις ταλικές τράπεζες, πρώτα απ' όλα Θέλω να σας πω ότι μεταξύ της προηγούμενης εβδομάδα και σήμερα η οικονομική κατάσταση των τραπεζών αυτών δεν έχει αλλάξει. Έγινε μια ψηφοφορία πολιτική, η οποία άλλαξε κάπως την κατάσταση, αλλά εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν λύσεις στις διάφορες καταστάσεις. Οι λύσεις αυτές μπορεί να πάρουν χρόνο και όπως είπα και πριν, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι καθορισμένοι κυρίως στο BRT, στο SSM, στον νεοκοπτικό μηχανισμό και αναφέρεται και στην ανακαίωση της Digicom. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω από αυτού. Στην περίπτωση ε, προληπτικής ανακεφαλοποίησης, τότε παρεμβαίνει ο SSM. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. and Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την κυρία Κένινγκ για τόσα μας είπε σήμερα το απόγευμα. Εδώ είμαι. Είμαι από την Ιρλανδία. Και είδα τι έγινε με το bailout για τις Ιρλανδικές τράπεζες. Πολύ χάρηκα που την άκουσα να λέω ότι οι κανόνες είναι κανόνες, ότι έχουμε κάνει βήματα ιστορικά από το σύστημα bailout στο σύστημα bail-in διάσωση με ίδια μέσα. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και χαίρομαι που το είπε έτσι ξεκάθαρα και δυνατά για να το ακούσουμε όλοι. Οι ερωτήσεις μου τώρα σε σχέση με το ενίο Συμβούλιο Εξηγένσης. 10 ε, δις, είχαμε πει σε 8 χρόνια 25 δις, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό για την πρώτη μου ερώτηση. Επειδή απάντησε και στον κύριο Νταμάσης νωρίτερα, για το χώρα προς χώρα, μπορεί να απαντήσει και τράπεζα με τράπεζα ότι θα γίνει η διαδικασία. 1,8 δις έβαλε η Ιρλανδία από τον Ιρλανδικό τραπεζικό ε, τομέα. Δεν ξέρω αν το έχει συζητήσει με τις εθνικές τράπεζες. Κάτι ακόμα για τη συνεργασία που θέλει και που πετυχαίνει το νέο Συμβούλιο Εξυγένση για να υπάρχει μια υποπτική προσέγγιση στο σύστημα. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αν ναι, πού. Ώστε να υπάρχει διάλογος με τις εθνικές αντίστοιχες εποπτικές αρχές. Και τέλος σε κάτι που ρώτησαν και άλλοι για τα MRLs. 8 με 10 χώρες μέλη έχουν ε, τράπεζες με 5%. Θα πρέπει τα κακά δάνεια. Γι' αυτό θα πρέπει και εκείνη να μας πει τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στη, στον τραπεζικό τομέα συνολικά, γιατί μπορεί να μεταδοθεί το φαινόμενο. Απάντηση, ευχαριστώ. Θα αρχίσω με το Ταμείο. Τα 55 δις υπολογίστηκαν από την αρχή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποθέτοντας ότι πρόκειται για 1% των αγαλημένων ε, αποζημιώσεων αυτή την περίοδο. Αν δούμε τα σημερινά νούμερα, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα νούμερο που να είναι περισσότερο από τα 55 δισεκατομμύρια. Προς το παρόν, και σε όσους αρέσουν τα μαθηματικά μπορούν να το φανταστούν, το ταμείο αυτό πρέπει να φτιαχτεί βήμα-βήμα για τα 8 πρώτα χρόνια για να φτάσει στο 1% στο τέλος. Βέβαια το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα είναι μετά από 8 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και πέρσι αποφασίσαμε να έχουμε μια συνεισφορά που είναι 1,05% των περσινών καταθέσεων υποθέτοντας ότι θα υπάρξει αύξηση που θα μας οδηγήσει σε 65 ίσως δις. Δεν ξέρουμε, το προσαρμόζουμε βήμα-βήμα. Εγώ δεν βλέπω κανένα επιχείρημα, αλλά δεν έχω και τα νούμερα μπροστά μου, για την Ιρλανδική εισφορά, κατά πόσο αυτή θα αλλάξει. Αυτό που βλέπουμε, και ισχύει κυρίως για την Ιρλανδία, ότι η μετακίνηση τραπεζών ε, εντός και εκτός μιας χώρας αλλάζει τη βάση. Οπότε θα αλλάξει τότε και η ετήσια συνεισφορά. Αλλά εδώ κάνουμε ίση μεταχείριση. Έρχομαι στη δεύτερη ερώτησή σας. Συνεργασία με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που για μας είναι ο κατεξοχήν ε, εποπτικός ε, φορέας. Και υπάρχει ένας τομέας που πάντα αναφέρω, Η πιο εύκολη απώλεια είναι η πρώτη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να φροντίσουμε προχωρώντας και το συνειδητοποιούμε όλοι είναι ότι μέτρα έγκαιρης παρέμβασης πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς έγκαιρα, νωρίς και όχι στις 12 και 5. Και αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ήπιο τρόπο. Δεν υπάρχει όμως διαφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ' αυτού και έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ μας. Τέλος, NPS, επ' αυτού το κοιτάμε όχι μόνο σε μία μόνο χώρα, όταν εξετάζουμε την μία την άλλη κατάσταση, Εντάξει, μπορεί να είναι μεμονωμένη μία ή άλλη κατάσταση, οπότε μπορείτε να προβλέψετε τι θα κάνετε για τη μεμονωμένη περίπτωση. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Όταν έχουμε να κάνουμε με σχέδια εξυγίανσης, πάντα έχουμε την ερώτηση πώς θα αντιδρούσατε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση τράπεζας. Πάντως, πάνω απ' όλα, συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να επιτεχυνθεί το έργο των MPLs. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Κόνιχ, για τα όσα μας εκθέσατε. Απόψε. Δύο πράγματα μας είπατε σε αυτή τη συζήτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αφενός με σαφήνεια είπατε ότι Διαφορετικά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς λέτε ότι σε σχέση με μια χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να θεωρείται ως ένα καθαρό paybox, ως ένας κουμπαράς. Έχει κάτι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, διότι έχει διαφορετική άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, είπατε ότι εναλλακτικά μέτρα, alternative measures, πρέπει να είναι εφικτά και δυνατά. Και είπατε και κάτι τρίτο πολύ ενδιαφέρον, ότι στα εναλλακτικά μέτρα όχι μόνο πρόκειται για μέτρα ε, ε, τόνωσης ή ενδυνάμωσης των θεσμών, θεσμικών οργάνων, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Και αυτό περισσότερο είναι η κατανό, περισσοτερο και αυτο περισσοτερο ειναι η κατανοηση για τα νομοθετικά πράγματα τα οποία απαιτείται να υπάρχει σήμερα. Και έτσι λοιπόν δώσατε και ένα παράδειγμα και είπατε εναλλακτικά μέτρα. Για παράδειγμα, σχέση των ε, πελατών με λογαριασμούς που μπορεί να μεταφέρονται σε άλλη τράπεζα. Αν αυτό είναι κάτι πιο ευνοϊκό από μια καθαρά εξηγιαντική δράση, ότι δηλαδή οι πελάτες ε, με ένα τέτοιο μέτρο βοηθούνται πολύ περισσότερο από ότι με μια δράση κουμπαρά. Διότι το γενικό όφελος τονώνεται το δημόσιο όφελος, διότι υπάρχει μικρότερη δαπάνη που συνεπάγεται αυτό το μέτρο. Και για τη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, ίσως αυτό μπορείτε να μας το επεξηγήσετε περισσότερο. Πώς κάτι τέτοιο λειτουργεί, ε, ειδικά και εξειδικευμένα, διότι δεν είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αυτό το μέτρο. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το backstop, δηλαδή τη δυνατότητα να πάψει η διαρροή. Όταν έχει πλέον απαντληθεί το χρήμα και δεν υπάρχει διότι διαφορετικά χάνουν όλη την αξιοπιστία ε, σε μια τράπεζα. Παράδειγμα για τον εξευρω... εξευρωπαϊσμό τέτοιων ε, ε, δεξαμενών δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει μια σφραγίδα που θα θέτει τέρμα στην απάντηση χρήματος από μια τέτοια δεξαμενή ώστε για παράδειγμα υπό την μορφή ρητρών που θα μπορούσαν να ενταχθούν μέσα σε τέτοιου είδους μέτρα. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτα την πρώτη ερώτηση. Όταν ανέφερα το DGF και τα εναλλακτικά μέτρα, αναφερόμουν ουσιαστικά στο FDIC. Για την τελευταία δεκαετία χρησιμοποίησε εναλλακτικά μέτρα, δηλαδή μεταφορές όσον αφορά πελάτες προς ένα άλλο θεσμικό, πελατών προς ένα άλλο θεσμικό όργανο και εντάσσοντας ε, το ε, όργανο αυτό σε διαδικασίες ε, αφαιρεγγιότητας για την εξυγίανση. Έτσι λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο υλοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη και έχετε δίκιο ότι δεν αποτελεί τμήμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου θα είχαμε ένα είδος κουμπαρά από την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ε, επανεξετάζεται όχι ως μια ανοιχτή επιταγή, αλλά εξετάζοντας και τα εναλλακτικά μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιούν τον στόχο να μην είναι περισσότερο δαπανηρά από ότι ε, μια διαδικασία κουμπαρά για την αντιμετώπιση αφαιρεγγιότητας. Και εμεί είπαμε ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν μια πιο λειτουργική λύση και πρόταση και αυτή ήταν η τοποθέτησή μας ευθύς εξ αρχής για το, τη δυνατότητα σφραγίδας ε, επιτέλους ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας ότι ολοκληρώνεται μια διαδικασία ε, όπου και ε, οι εκκρεμότητες ε, ρυθμίζονται, η χώρα που έχει την αρμόδια υπεύθυνη κυβέρνηση μπορεί να επιταχύνει. Όταν κάνουμε λόγο για μια τέτοια σφραγίδα που τίθεται, δεν γίνεται λόγος για μια ανοιχτή διαδικασία. Πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο πρέπει να μπορεί να ε, αποσβαίνεται μέσω εισφορών που θα καταβάλλονται προς ένα θεσμό, σε ένα θεσμικό όργανο. Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε κάτι τέτοιο. Αν στο ευρωπαϊκό επίπεδο προτινόταν να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Αλλά επικεντρωνόμαστε στο Ταμείο Εξυγίανσης και εφόσον επιθυμούν να υλοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη είμαστε σε ετοιμότητα να έρθουμε ως αρρωγή και να βοηθήσουμε. Μα το παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας για την χρηματοδότηση και γιατί σας ρωτάω. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες τελικά τιμωρούνται σε σχέση, σε σύγκριση με τις Αμερικανικές τράπεζες εξαιτία της Βασιλείας 3, που εφαρμόστε σε όλες τις τράπεζες στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ μόνο στις μεγάλες τράπεζες. Και αυτή είναι μια διαφοροποιημένη μεταχείριση και θέλω να ξέρω τη γνώμη σας από αυτού. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι τιμωρούνται κάποιες τράπεζες, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες μεταχειρίζονται διαφορετικά τις δικές τους μικρές ε, τράπεζες. Διαφάνεια ε, από ταμιεύσεις έχουν ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο για αυτές. Ενώ η δική μας και οι κανόνες που βγαίνουν από την Επιτροπή Βασίλης είναι μόνο για τις μεγάλες τράπεζες και είναι δύσκολο βέβαια να καθορίσει κανείς τη διαχωριστική γραμμή. Αυτό οδηγεί σε τεράστια διαφοροποίηση σε επίπεδο λεπτομεριών, ναι. Κατά πόσο είναι σε δυσμενή θέση δεν ξέρω, δεν, δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί εξαρτάται αναπερίπτωση. Σίγουρα θα έπρεπε να δούμε την αναλλαγικότητα και τα λοιπά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλφρετ Σάντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα προγράμματά σας ε, για το 2017 δίνεται προτεραιότητα ε, στο να υπάρξει κάποια ιεράρχηση των προγραμμάτων εξυγίανσης. Επίσης, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εναρμόνιση των εθνικών της εθνικής νομοθεσίας και λέτε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο περιθώριο για εναρμόνιση. Συμφωνείτε ότι αν ακολουθήσει κανείς αυτή την προσέγγιση υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει σε μια μαϊκή συνταγή για όλα. Ξέρω ότι θα πείτε όχι, αλλά θέλω να ρωτήσω τι μπορεί κανείς να κάνει για να αναχαιτήσει αυτό το πρόβλημα, κυρίως όταν, έχει, όταν πρόκειται για ε, μεσαίες κεφαλαιοποίησεις ε, τράπεζας. Δεν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούν τελείως διαφορετική ε, μεταχείριση. Οι μηχανισμοί, ε, εφαρμοσμένοι μηχανισμοί που έχουν αρμονιστεί θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να περιοριστεί η χρηματοπιστωτική ευελιξία σε ένα αρκετά μεγάλο, μικρό περιβάλλον και οι μικρές τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Δεν υπάρχει λοιπόν σε γενικές γραμμές η δυνατότητα οι διαδικασίες εναρμόνισης να προάγουν περαιτέρω την, ε, τον ολιγοπολιακό χαρακτήρα των ε, τραπεζών. Αυτό θέλετε όταν μιλάμε για benchmarking, ε, κατ' ουσίαν ε, μπαίνουμε σε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε κάποιες τράπεζες ε, όπου οι ομάδες μας, οι συνεργάτες μας, έχουν εντοπίσει πολλές ε, λειτουργίες και μετά έχουμε τράπεζες που είναι μεγαλύτερες και έχει κανείς ε, εντοπίσει τρεις-τέσσερις λειτουργίες. Όταν μιλάμε για benchmarking ε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούμε τα κριτήρια όταν ορίζουμε το τι είναι κρίσιμο σε κάθε μία από τις ομάδες μας. Δηλαδή όταν ορίζουμε το πόσο σοβαροί θέλουμε να είμαστε, να έχουμε τα ίδια κριτήρια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και εδώ δεν συμμερίζομαι την άποψή σας ε, για το διαχωρισμό ανάμεσα στο βορρά και τον νότο. Έχουμε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα γιατί υπάρχουν ε, Ινστιτούτα τα οποία ε, χρηματοδοτούνται τελείως διαφορετικά, δηλαδή έχουν μετοχικό κεφάλαιο, έχουν καταθέσεις και μετά υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά υπάρχουν στην Ευρώπη και στον Βορρά και στο Νότο και αυτά είναι τελείως διαφορετικά από επενδυτικές τράπεζες. Πρέπει λοιπόν κανείς να τα εξετάζει αυτά διαφορετικά και ενδέχεται να καταλήξει και σε διαφορετικές σκέψεις. Όμως για μας ε, benchmarking είναι απαραίτητο διότι ακολουθούμε και τη γραμμή όπου έχουμε συγχώνευση τραπεζών σε διάφορες χώρες, δηλαδή δεν θέλουμε να συμπεριφερθούμε σε μια χώρα διαφορετικά από ό,τι σε μια άλλη. Και όταν μιλάμε για εθνικής φύσεως θέματα, υπάρχει ένα παράδειγμα που έχουμε διαπιστώσει, δηλαδή λόγω ε, των ε, λεπτομερών ε, νομοθετικών διατάξεων για την αφεργιότητα, οι τράπεζες καλούνται ε, να συστήσουν μια holding εταιρεία. Αυτό μπορεί να μην ισχύει σε άλλες χώρες ή για να το πω αλλιώς, ξεκινάμε με πρόγραμμα εξυγίανσης και αυτό μετά πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να προσαρμοστούμε στο εθνικό δίκαιο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες όχι με μαγικές συνταγές που είναι ισχύουν για όλους, αλλά να υπάρχει μια συνέπεια μέσα στην ε, Τραπεζική Ένωση. Νίνα Γκέι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας. Ένας άλλος βασικός στόχος του προτινόμενου παχέτου είναι να μεταφέρουμε το βάρος από τους φορολογούμενους στους πιστωτές και εγώ το στηρίζω αυτό. Αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει κάποιες πτυχές της πρότασης της Κομισιόν. Οι τράπεζες θα μπορούν να αξιολογήσουν μόνες τους κατά πόσον ε, θα έχουν 3,5% από το 18% ε, που να μην είναι subordinated και αν ισχύει αυτό ε, δεν ε, είναι παραμπίση της αρχής NCWO. Εγώ ανησυχώ γιατί η αρχή εξυγίανσης ε, δεν καταλήγει σε αυτή την απόφαση και αυτά εναπόκεινται στις τράπεζες. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό υπονομεύει το βασικό στόχο της πρότασης και από το δεύτερο που θέλω να πω είναι η πρόσβαση της Κομισιόν που ε, λέει ότι οι τράπεζες Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με το TLAC. Όμως, ε, αυτό θα μπορούσε να αφορά και τις ε, συστημικές τράπεζες. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος ε, όσο έχουν τώρα τα πράγματα να έρθει κανείς αντιμέτωπος με τους κανόνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Κοιτάξτε, ε, ανησυχώ λιγάκι αν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η τράπεζα εκείνη η οποία αποφασίζει κατά πόσον το 13,5% αρκεί ως υποκείμενο, το πούμε, χρέος. Αυτό το κάνει η Κομισιόν. Ε, υπάρχουν οι ε, ευρωπαϊκές εξαιρέσεις, αλλά έχετε απόλυτα δίκιο ότι αυτό πρέπει να μετράτε και η αρχή της ε, εξυγίανσης καλείται εδώ να παρέμβει. Διότι Αυτά ισχύουν μόνο εφόσον η τράπεζα πραγματικά μπορεί να εξηγεντεί ε, χωρίς να ζημιωθεί χειρότερα κανένας πιστωτής. Και πάμε σε μια άλλη συζήτηση σχετικά με την ιεράρχηση των ε, πιστωτών. Ε, κατά την άποψή μου λοιπόν αυτό ισχύει για την αρχή εξυγίανσης. Εκείνη θα αποφασίσει και όχι η τράπεζα. Η δεύτερη ερώτηση που κάνατε, κατά πόσον οι απαιτήσει για τις ενδιάμεσες εταιρείε holding. Εγώ δεν θα έλεγα ότι αυτό ε, στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το ζητάνε και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Προς το παρόν είναι μια έννοια η οποία θα πρέπει να διευκολύνει τη δυνατότητα αυτών των τραπεζών να εξηγενθούν στην Ευρώπη και βεβαίως μετά ε, πρέπει να δούμε τις ε, λεπτομέρειες. Ανέκαθεν ήμουνα κατά της πρότασης ε, των ΗΠΑ να υπάρχει μια ενδιάμεση holding εταιρεία. το ΤΙΛΕΚ e είναι ένα είδος περιχαρακόμματος αλλά είναι και ένα κομμάτι μιας ε, έννοιας όπου πρέπει κανείς ε, να διασφαλίσει είτε είναι MRL είτε το ΤΙΛΕΚ e θα πρέπει να εντάσσονται σε μεγαλύτερες ε, μονάδες εξυγίανσης. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες άλλες ενέργειες, αλλά για μένα όλα αυτά είναι λογικά. Ευχαριστούμε. Η Ντανούτα, έτοιμη για την ερώτησή σας. Ναι, ήμουν στην άλλη επιτροπή που είμαι εγώ ο πρόεδρος και δεν μπόρεσα γι' αυτό να έρθω νωρίτερα. Ελπίζω κύριε Κένιγκ να μην σας ρώτησαν για το CCP ήδη. Θέλω να σας πω ότι αυτή η νέα πρόταση που πήραμε από την Επιτροπή προβλέπει μια κατάσταση για καθάριση μεγάλης τράπεζας. Αν υπάρχει λοιπόν τέτοια περίπτωση όπου μια μεγάλη τράπεζα ε, βρεθεί σε δυσκολία την ε, BRD, την οδηγία, υπάρχουν διατάξεις για τέτοιες περιπτώσεις. Εσείς όμως πώς θα λάβετε υπόψη σας στην πράξη τέτοιου είδους συνεργασία όσον αφορά την εξυγίανση. Δεν θα είναι το CCP που θα πληρώσει υπερβολικά για τα λάθη που έχουν κάνει οι τράπεζες, αν μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο δηλαδή ανάμεσα στις ε, δικές σας αρμοδιότητες και του CCP. Προς το παρόν, εμείς, το δικό μας ενίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, δεν έχει τίποτα κοινό με το CCP. Με μία εξαίρεση ότι κάποια CCP έχουν άδεια για τραπεζικές δραστηριότητες, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά γενικώ η εξυγίαση CCC δεν είναι χαρτογραφημένη δραστηριότητα, όχι μόνο στην Ευρώπη, ούτε κι αλλού. Μερικές φορές το βράδυ πηγαίνω στο steering committee και πιέζουμε σε διεθνές επίπεδο ακριβώς για να πούμε ότι οι ρυθμιστές, οι νομοθέτες έκαναν το σύστημα CCP όπως το έκαναν για πολύ ξεκάθαρο τρόπο, γιατί τα προϊόντα τους έτσι χαίρουν περισσότερης διαφάνειας και άρα υπάρχει μεγαλύτερη αντοχή στις κρίσεις. Αλλά βέβαια όλοι πρέπει να ξέρουμε τι είναι. Και το βασικό σενάριο είναι ότι ένα ή δύο από τα μεγαλύτερα μέλη clearing δεν τα καταφέρνουν και οι θέσεις τους δεν μπορούν να κλείσουν όπως περιμένουμε. Παγκοσμίω οι περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις είναι G-SIPs και όχι μόνο σε ένα CCP αλλά σε πολλά τέτοια. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αλυσιδωτή κατάσταση που ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ. Θα έπρεπε όμως να καθορίσουμε σε ποιο σημείο παρεμβαίνουμε και τότε όντω θα παρέμβουμε γιατί τα g που είναι δικιά μας αρμοδιότητα ή θα είναι αυτοί που δεν θα τα έχουν καταφέρει ή θα είναι αυτοί οι οποίοι εν δυνάμει θα έχουν απώλειες εξαιτίας της αποτυχίας κάποιου CCP. Για όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε πού καταλήγουν αυτές οι απώλειες. Και αυτό είναι που έχει στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι που συζητιέται εκ παραλλήλου σε διεθνές επίπεδο. Αν είμαστε αρκετά έξυπνοι, θα καταλήξουμε να έχουμε παράλληλες καταστάσεις και όχι τη μία που να κυριαρχεί της άλλης. Αυτό συζητιέται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άφησε ανοιχτά κάποια σημεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν έχω άλλον ομιλητή ή έχω. Ωραία. Σβέν, παρακαλώ. Μόνο για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είχα ρωτήσει προηγούμενα λόγω χρόνου δεν καταφέρατε φαντάζομαι να, απαντήσω, να απαντήσετε την διάσταση όσον αφορά τις τρίτες χώρες σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Από ό,τι γνωρίζω η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά ανοίγει μια θύρα, μια δυνατότητα, ότι δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν bail-in ρήτρε σε χρηματοοικονομικά μέτρα και μέσα όσον αφορά τρίτες χώρες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση επ' αυτού. Δεν είναι μάλλον μια πρόσκληση ώστε να υπάρξουν τέτοιου είδους ε, ε, προτερήματα και προνόμια εκτός Ευρώπης ε, για τέτοιου είδους κινήσεις διότι μάλλον ε, ίσως ε, μπορεί να εκπλήσει κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως αλλαγή σε σχέση με την πρόταση όπως είχε προταθεί και θα θέλαμε να ακούσουμε ποια είναι η δική σας άποψη από αυτό. Πράγματι, ε, με παραξένεψε. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στο άρθρο 55 και στο άρθρο 55 νομίζω απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Η δική μου η προσέγγιση είναι και πάλι εδώ υπησερχόμεθα σε πολλές λεπτομέρειες γραμμή αναγραμμή. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση από ό,τι γνωρίζω όσον αφορά το μη εφικτό και ίσως και την μη ύπαρξη ανάγκης να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια μιας σύμβασης σε μια τρίτη χώρα, ενώ ο κανονισμός ήταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ενέτασε πολλά θέματα σε αυτόν. Και εδώ για μία εξαίρεση de και όχι τίποτα άλλο, αν διατυπωθεί με αυτόν τον τρόπο και θα πρέπει να εξεταστεί η διατύπωση για άλλη μία φορά, τότε είμαστε υπέρ μίας ε, εξαίρεσης de γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ε, πηγαίνουμε από πρόσκομα σε εξυγίανση αλλά αν ήταν κάτι παραπάνω ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο για κάτι τέτοιο. Ελπίζω ότι απαντώ επί της παρατήρησής σας. Ε, υπήρξαν κάποιες ανησυχίες που διατυπώθηκαν και γι' αυτό ζήτησα να επανεξεταστεί. Θα θεωρούσα ότι ο κανονισμός, ο κανόνας de θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένος. Εδώ όμως δεν υπάρχει χρονικός ε, περιορισμός και λέγεται αν νομικά ή δομικά, διαθροτικά μπορεί να μην ε, είναι κάτι τέτοιο εφικτό, το κατανοώ αυτό, αλλά αυτό θεωρείται σαν μια δυνατότητα δράσης. Ε, ενώ όταν έχουμε μια αρχή η οποία θα πρέπει να δεσμεύει τις δράσεις μας, ε, δεν θα πρέπει μέσω τέτοιων δράσεων να δεσμευόμεθα το de minimis, η ρύθμιση de minimis νομίζω θα είχε κάποιο νόημα αν ήταν σε αυτό το πλαίσιο μόνο. Η πρόθεση είναι να υπάρχει μια εξαίρεση de minimis, των προδιαγραφών. Ρωτήστε όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εκείνοι συνέταξαν την πρόταση. Εγώ απλώς την ερμηνεύω. Ναι, γι' αυτό τον λόγο το επανεξετάζω κι εγώ. Ναι και πράγματι από πλευράς ε, νομοθετών θα πρέπει αυτό να εξετάζεται ως ε, έργο. Υπάρχει μια ευκαιρία εδώ λοιπόν σε σχέση με την εξέταση αυτής της ερώτησης και αυτό το οποίο εσείς υπενηχθήκατε σε σχέση με τις ε, προκλήσεις που θα πρέπει να βοηθηθούμε να αντιμετωπίζονται σε σχέση με τρίτες χώρες. Εσείς αναφέρεστε σε σχέση με την ελαστικότητα όσον αφορά την ιεραρχική ένταξη αυτών των θεμάτων μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ή τι είναι αυτό το οποίο εσείς στοχεύατε να πείτε. Ποια είναι η δική σας άποψη, μπορείτε να μας την επεξηγήσετε. Ε, σίγουρα κάποιος βαθμός δεν θα το αποκαλούσα ευελιξίας, αλλά εξέτασης μιας στρατηγικής εξυγίανσης σε σχέση με ένα ε, θεσμικό όργανο ε, ή ταμείο σε σχέση με ένα τραπεζικό ε, φορέα, αλλά αυτό το οποίο αναφερόμουν πιο εξειδικευμένα είναι ο χρονικός παράγοντας. Δεν δώσαμε κάποια χρονική διάρκεια ή ε, περιορισμό, αλλά όταν υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα χρειάζεται σαφώς περισσότερος χρόνος για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο μείζο πρόβλημα. Όμως ένας μεγάλος βαθμός αυτών που ταυτοποιήσαμε, αν υιοθετηθεί η πρώτη προσέγγιση που αφορά πολύ μικρότερο αριθμό από εκείνο, από τον αριθμό που αναφέρεται, από 70 τράπεζες θα όταν αναφέρεται ότι έχουμε περίπου 120, 100 ή 120 δις, αλλά όχι τα 700-800 δις τα οποία είχαν ε, αναφερθεί και είχαν τέθει σε κυκλοφορία ως υποθέσεις. Αλλά αυτό ένα παράδειγμα. Αυτό το ποσό το οποίο συσχετίζεται με το γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί από διαφορετικής πλευράς ε, επιλέξιμο ή μπορεί να υιοθετηθεί μια πιο αυστηρή προσέγγιση με την δομημένη προσέγγιση όσον αφορά την ε, ε, τις ασφάλειες ε, που θα έπρεπε να δημιουργηθούν ή και τη διπλή μόχλευση στη Γερμανία έναντι της προσέγγισης των ΗΠΑ, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταποκρίνεται περισσότερο και δημιουργεί ένα τέτοιο μεγαλύτερο περιθώριο, πράγμα το οποίο θα μας έδινε την ευκαιρία να εκτάσουμε τις θετικές δυνατότητες. Το λέω για να σας δείξω ότι δεν, έχουμε, είμαστε θεσμικά ανέστητοι επ' αυτού και δεν το αγνοούμε και θα επανέλθουμε σε σχέση με το χρονικό όριο η διάρκεια. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ θετική και γόνιμη αυτή η καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων, δύσκολες ερωτήσεις, ισορροπημένες περιεκτικές απαντήσεις και μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας τώρα. Η επόμενη την Πέμπτη στις 9 με σημαντικές ψηφοφορίες που θα διεξαχθούν για την securitization και θα έχουμε και μια κοινή συνεδρίαση, ναι το επαναλαμβάνω, θα ψηφίσουμε Econ Libe συνεδρίαση, σε Econ συνεδρίαση και σε σχέση με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξη κατά του πλησίματος χρήματος. Σας ευχαριστώ για το ότι είσαστε παρούσες και παρόντες και προσβλέπουμε στην επόμενη τέτοια ακρόαση. Ευχαριστώ. Γεια σας.